Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Έχουμε φτάσει σίγουρα στο σημείο 16. Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Έκθεση του κυρίου Φιέλνερ, την οποία σκοπεύουμε να ψηφίσουμε την επόμενη φορά που θα συνεδριάσει η Επιτροπή μας. Α, να ακούσουμε πότε θα ψηφιστεί. Αφού δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στον εισηγητή για να μας ενημερώσει, να μας εισαγάγει και πάλι στο θέμα. Κύριε Φιέλνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ξανασυζητήσει για την έκθεση αυτή ε, στο παρελθόν και τώρα καλούμαστε να συζητήσουμε τις τροπολογίες που είναι πάνω από 300 παρακαλώ στον αριθμό και μπορεί κανείς να θεωρεί ότι πώς να το πω ότι με έχουν κατακλείσει τροπολογίες και έχω πελαγώσει. Όχι. Τις έχω διαβάσει, τις έχω μελετήσει και ε, νομίζω ότι πολλές πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Από τις 300 αυτές τροπολογίες έχουμε πολύ μεγάλη συμφωνία. Σε πολλές. Εγώ έδειξα πνεύμα συνεργασία. Το είχα πει και από την αρχή κιόλα. Το είχα δηλώσει ότι ελπίζω να καταθέσετε ε, πολλέ τροπολογίε, όπω και για το. Και πολλέ με βρίσκουν σύμφωνο. Θα πρέπει να χρειαστούν πολλοί συμβιβασμοί που δεν θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Οι πρώτες τροπολογίες δεν μ' αρέσουν ε, γιατί είναι τροπολογίε που θέλουν να καταρρύψουν ολόκληρη την πρόταση, να την ακυρώσουν. Όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βρούμε μια συμφωνία για το θέμα αυτό και όχι να απορρίπτουμε συλλήβδιν την πρόταση. Αλλά γενικά είναι περισσότερες οι ε, συμφωνίες στα θέματα που μας ενώνουν από εκείνα που μας χωρίζουν. Τι θέλουμε λοιπόν εμεί, τι είδου πληροφόρηση πώς θα πρέπει να ενημερώνεται το κοινό από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ε, εδώ μιλώ για τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία του φαρμάκου, ε, για τις δόσεις, ε, για γενικές πληροφορίες ιατρικής φύσης. Σε αυτό συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές και να κοινοποιούνται μετά ε, θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στο σύστημα push και pull, δηλαδή να παρέχεται η πληροφορία ή να την αναζητάει κάποιος. Αυτό το push, δηλαδή που είναι ε, μια πληροφόρηση που δίνει η εταιρεία, να αφορά μόνο ιατρικά έντυπα και να μην ενημερώνεται το ευρύ κοινό. Να απαγορευτεί αυτό ζητούν ορισμένοι και ε, άλλοι θέλουν να αλλάξουν τη διατύπωση ε, από διάδοση της προφορίας σε πρόσβαση στις προφορίες. Δηλαδή όταν θέλει κάποιος μια προφόρηση να την ε, ψάχνει. Και... Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει μια στοιχειώδης προφόρηση να παρέχεται χωρίς να χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος ασθενή να την αναζητήσει. Επίσης, τίθενται και διάφορα ζητήματα έγκρισης και αδειοδότησης ε, πριν ε, προχωρήσουν σε διάφορες ενέργειες οι φαρμακοβιομηχανίες. Άλλο θέμα είναι τα διάφορα ε, φυλάδια ακριβώ που βρίσκουμε μέσα στα φάρμακα. Δεν είναι ομοιόμορφα, δεν είναι τυποποιημένα, είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα και πολλές φορές δυσανάγνωστα. Ε, σε πολλές ε, περιπτώσεις, ε, σε διάφορες ενημερωτικές εκστρατείες, χάνουν το στόχο τους και παραπληροφορούν και παραπλανούν και οδηγούν σε ανασφάλεια. Άλλες τροπολογίες που υποστηρίζω εγώ και είναι ενδιαφέρουσες, είναι κάπως διαφορετικές από την αρχική πρόταση και πρόκειται για ακριβώς την αλλαγή των οδηγιών μέσα στα φάρμακα. Τα κράτη-μέλη όμως ε, είναι αρμόδια για αυτό το θέμα και ε, οι διάφοροι οργανισμοί φαρμάκων. Δεν θα πρέπει να τα κάνει όλα η φαρμακευτική εταιρεία. Σα είπα λοιπόν υπάρχουν πολλές τροπολογίε, ε, πολλές συμφωνώ γιατί πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και είναι και οι περισσότερε άλλωστε σε όλο. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμού. Εύκολο δεν θα είναι, θα χρειαστεί χρόνο, γι' αυτό θα πρότεινα να μην ψηφίσουμε την επόμενη φορά γιατί χρειάζομαι χρόνο. Καταλαβαίνετε, για 300 τροπολογίες χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να καταλήξω σε συμβιβασμούς. Ε, αυτές ήταν οι τροπολογίες στις οποίες συμφωνώ. Τώρα έρχομαι σε κάποια θέματα που είναι κάπως δύσκολα και ακαθόδη, δεν απέχουμε και τόσο πολύ, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε τεχνικές φωνίες. Ήταν κάποια θέματα πάρα πολύ επίμαχα που συζητήσαμε με τους ε, συναδέλφους για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Δεν συμφωνούμε εκεί σε όλα. Θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέλφους. Ακριβώς για τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις κεφασίες των φαρμάκων θέλω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Το ξέρω ότι είναι τεχνικό το θέμα. Δεν ξέρω θα πρέπει να υπάρχει κεντρική διαδικασία που να τα ρυθμίζει όλα αυτά. Και μετά υπάρχει ένας τρίτος ε, τομέας, μια τρίτη ενότητα τροπολογιών που αφορούν το διαδίκτυο. Ότι αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει μόνο, δεν συμφωνώ. Να σας πω τι συμβαίνει στη Σουηδία. Μπορεί κανείς να ζητήσει τις προφορίες αυτές, να τις παραγγείλει. Γιατί δεν έχει όλος ο κόσμος διαδίκτυο. Και ε, μπορεί λοιπόν να παραγγείλει αυτή την πληροφόρηση και να τη λάβει ταχυδρομικός ή ας πούμε η τυφλή ακόμα και σε γλώσσα μπράιε Δεν θα πρέπει ε, λοιπόν να είμαστε προσκολλημένοι υπερβολικά στο διαδίκτυο. Ε, για τους ελέγχους είναι ίσως το πιο δύσκολο. Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι, πώς θα ελέγχονται αυτές οι πληροφορίες που δίδουν οι εταιρείες για τα φάρμακα. Ορισμένοι ε, λέγουν ε, να τα αναλάβουν αυτά οι υγειονομικές υπηρεσίες ή ε, οι οργανισμοί φαρμάκων. Υπάρχουν αφενός ουσίες οι οποίες έχουν εγκριθεί, κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά κάποιες χώρες έχουν προβλήματα μέχρι και συνταγματικής φύσεως σε ό,τι αφορά τον πρώτερο έλεγχο ουσιών που κυκλοφορούν στη χώρα πριν κυκλοφορήσουν. Δεν θα πρέπει όμως να παρέχετε ενημέρωση για ουσίες που δεν κυκλοφορούν ακόμα στο εμπόριο γιατί δεν έχουν ακόμα εγκριθεί στα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο τώρα Όταν θέλει μια εταιρεία να ενημερώνει για ένα φάρμακο, για μια ουσία, λέει ε, να περιορίζεται στη δική τη ιστοσελίδα. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Υπάρχουν φαρμακευτικές εταιρείε που συνεργάζονται, α πούμε, με κάποιε άλλε και έχουν ε, πληροφόρηση από διάφορε πηγέ. Στη ε, Σουηδία και πάλι, πώ έχει κατάσταση. Όλε αυτέ οι πληροφορίε βγαίνουν σε μια κοινή ιστοσελίδα για όλα τα φυλάδια τη συσκευασία των φαρμάκων. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται κάτι τέτοιο αλλά να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Τώρα, για διάφορες εκστρατείες για θέματα υγείας. Εκφράστηκε πολύ μεγάλη κριτική εδώ. Ε, πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει ε, να ρυθμίζονται σωστά αυτά τα πράγματα και ε, σε σχέση με σπάνιες ασθένειες ή ασυνήθιστες ασθένειες, γιατί κάποιο που μπορεί ε, να πάσχει από ένα πολύ σπάνιο ε, νόσημα, συγγνώμη, ε, να μην έχει καν στη χώρα του γιατρό που να είναι ειδικό για αυτή την ασθένεια. Ενώ η εταιρεία που βρίσκεται στην αιχμή της επιστημονικής καινοτομία μπορεί να τον ενημερώσει τον ασθενή για αυτή τη σπάνια ασθένεια. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται σε περίπτωση σπανίων νοσημάτων. Κάποιοι άλλοι λέγουν ότι θα πρέπει να απαγορεύονται τα βίντεο στο διαδίκτυο. Ναι, εντάξει, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση στο διαδίκτυο για φάρμακα, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θέλουμε τηλεοπτική ενημέρωση τύπου διαφήμισης, γι' αυτό θέλουν να το απαγορεύσουν οι συνάδελφοι το βίντεο. Και πάλι δεν είμαι τόσο απόλυτο εγώ. Θα μπορούσε να υπάρχει βίντεο να προβάλλεται στο διαδίκτυο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ένα φάρμακο. Να επιδεικνύεται αυτό σε βίντεο, να ξέρει ο στενής πώς θα το πάρει. Ας πούμε, μία ουσία ε, για την αντιμετώπιση του άσθματος ε, που ε, μπορεί να δείχνει το βίντεο πώς γίνονται οι σπνοές, πώς ε, θα πρέπει να παίρνει το φάρμακό του ασθενής. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν λέω ότι θα πρέπει όλες οι προφορίες για τα φάρμακα να γυρίζονται σε βίντεο και να βγαίνουν στο διαδίκτυο, αλλά όταν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, γιατί να απαγορεύεται, δεν το καταλαβαίνω. Αυτά προς το παρόν και είμαι βέβαιος ότι θα πούν και πολλά συνάδελφοι. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Πολλέ είναι και οι προτάσει. Καταλαβαίνετε τώρα πάνω από 300 τροπολογίες ε, πόσο ενδιαφέρον ε, έχουν οι συνάδελφοι. Πολλές τροπολογίες πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση όπως σας είπα, την οποία υποστηρίζω και εγώ στην έκθεσή μου. Κανονικά μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, να βρούμε μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε εσείς τι λέτε για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή Κρίστο Φέλνερ για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα το οποίο ε, προσελκύει την ε, προσοχή ε, των συναδέλφων όπως το αποδειχνεί ο αριθμός των τροπολογιών πρόκειται για την υγεία των ανθρώπων. Ως εκ τούτου ε, ο εισηγητής θεωρεί ότι για την βιομηχανία το θέμα αυτό είναι απλούστατα ένα μέσο για κάποιο σκοπό ουσιαστικά δηλαδή αυτός σκοπός και πρέπει να εξετάσουμε πώς πόσο, είναι, ε, ε, πόσο επιτρέπονται και πόσο πρέπει να εμποδίζονται και όχι μόνο για εμπορικούς λόγους διότι όταν ε, κάτι πάει στραβά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι και ξεκινάμε με τον Τζιλ Παρνιό σαν συντονιστή Σκιώδη. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Όπως το είπατε, όντως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα για τον 21ο αιώνα, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Όσον αφορά τους Ευρωπαίους, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή της, ε, του έτους 2010 να μπορέσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό όσον αφορά αυτές τις τις πληροφορίες. Δεν είμαστε στα πρώτα μας βήματα διότι ήδη το 2003 η Επιτροπή είχε αναφερθεί σε αυτήν την πληροφόρηση των ασθενών και είχε ζητήσει μαζικά να απορριφθεί η ε, ε, άδεια να χορηγούνται τα ε, φάρμακα ελεύθερα εάν πρόκειτο για φάρμακα βιομηχανιών που θα έπρεπε να συνταγογραφούνται. Δηλαδή ήδη τότε είχαμε εξετάσει πώς μπορούμε να ενημερώνουμε άμεσα τους ασθενείς. Διαβάζοντας λοιπόν αυτή την πρόταση οδηγίας και ιδίως σε σχέση με τον εισηγητή νομίζω ότι η οδηγία αυτή την οποία μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και αυτή η πρόταση κατά τη γνώμη μας ανοίγει την πόρτα για την άμεση προώθηση από τις εταιρείε, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Το μοναδικό κίνητρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αλλάξει αυτή η νομοθεσία είναι να εξυπηρετήσει τα φαρμακευτικά εργαστήρια ε, χωρίς όμως να καλύπτει τα συμφέροντα ούτε των κρατών μελών ούτε των ασθενών ε, και πρόκειται επιπρόσθετη γραφειοκρατία ε, και αύξηση των δαπανών και συνεπιφέρει και κίνδυνο για τους ασθενείς. Άρα κατά τη γνώμη μου προτείνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει τις προτάσεις αναθεωρήσεως και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μία επανεξέταξη του φακέλου όπως το είχε προτείνει τον Ιανουάριο ο Επίτροπος Ντάλη και αυτό για πέντε ουσιαστικούς λόγους οι οποίοι απαιτούν αυτή την επαναξιολόγηση της πληροφόρησης που δίνεται στους ασθενείς. Καταρχήν για να μπορέσει η Επιτροπή να σεβαστεί τη δημοκρατική διαδικασία διότι πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, βιομηχανικών εργαστηρίων και δεν έχει υπάρξει διαφάνεια στον τομέα. Πρέπει επίσης να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και ε, να προστατεύσουν τους πολίτες από την ε, άλογη χορήγηση φαρμάκων από την πύρα των Ηνωμένων Πολιτειών όπου η ελεύθερη συνταγογράφηση απεδείχθη εις βάρος των δημοσίων συμφερόντων. Πρέπει λοιπόν και εμείς να αποκομίσουμε τα συμπεράσματα των εμπειριών άλλων περιοχών. Συγχρόνως να συζητήσουμε με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών διότι υπάρχει υπάρχει μία αύξηση των δαπανών και το θέμα είναι πολιτικό. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν τους περιορισμένους πόρους για να ελέγχουν τα εργαστήρια των φαρμακοβιομηχανιών ή θα πρέπει να φροντίσουν οι ε, πολίτες να έχουν ανεξάρτητη και αντικειμενική πληροφόρηση και άλλωστε θα πρέπει να η Επιτροπή να επικεντρωθεί στους πραγματικούς στόχους που είναι να υπάρξουν νέα φάρμακα και όχι να ε, ε, δοθούν ε, άλλες πληροφορίες. Επίσης οι πολίτες πρέπει να έχουν ανεξάρτητη και ουσιαστική ενημέρωση και αξιόπιστη ενημέρωση όσον αφορά τα θέματα της υγείας τους για όλους αυτούς τους λόγους, τους πέντε ε, βασικούς λόγους που απαρίθμησα, πέραν των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, πιστεύω ότι σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναξιολογήσει την πρότασή της κατά τρόπον ώστε να ανταποκριθεί στις πέντε ανησυχίες τις οποίες διατύπωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πανιό για τους φιλελεύθερους ο, η κυρία Κράμερ έχει, ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Με συγχωρείτε, εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Χατζημαρκάκη που είναι συντονιστής, αλλά ευχαρίστω το πράτο διότι στην προηγούμενη θητεία ε, είχα εγώ τη θέση αυτή του σκιώδους ε, συντονιστή για το θέμα αυτό σκιώδη εισηγητή αλλά θα ήθελα να πω και μία φράση σχετικά με τον προλαλήσαντα α, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποπέμψουμε πλήρως την πρόταση αυτή πρέπει βέβαια α, θα πρέπει να απαγορεύσουμε ε, να προσφέρονται ε, εις τους πολίτες ε, ανεξέλεγκτες πληροφορίες. Αυτό όμως δεν έχει επιτευχθεί διότι βλέπουμε ότι πατώντας ένα κουμπί μπορεί ο καθένας να έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση εξαρτάται από την ξυπνάδα του, από τις τεχνικές δυνατότητες και από την περιέργεια των ατόμων ε, αν θέλουν αυτή την πληροφόρηση ή όχι. Οπότε είναι ε, παράλογο να λέμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε μία απαγόρευση που ισχύει από, από τα μέσα του προηγούμενου αιώνος. Εάν θέλουμε λοιπόν να περάσουμε αυτό το μήνυμα και αν επιμείνουμε ε, στην απαγόρευση οι ε, πολίτες δεν θα σωθούν και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά περιστατικά ασθενών μιλήσαμε τώρα για τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη στο στενό περιβάλλον πέντε ή έξι ε, πολίτες οι οποίοι παρόλη την απαγόρευση ε, έψαξαν αμφισβητούμενες πληροφορίες ε, στο διαδίκτυο, αγόρασαν τα φάρμακα και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Δηλαδή παρόλη την πλήρη απαγόρευση δεν μπορεί κανείς ε, να προστατεύσει τους ασθενείς από την παράπλευρη πληροφόρηση. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να βρούμε άλλες μεθόδους έχουμε τροπολογίες οι οποίες κατ' εμέ ε, είναι στη σωστή κατεύθυνση διότι προσπαθούν να διοχετεύσουν την πληροφόρηση σε οδούς στις οποίες οι ασθενείς θα ξέρουν ότι μπορεί κανείς να, έχουν, να έχει εμπιστοσύνη. Βέβαια χωρίς να υπάρχει πλήρη ασφάλεια. Οι τροπολογίες οι οποίες υπάρχουν ε, το τραπέζι που έχουν υπογραφεί από τον κύριο Χατζημαρκάκη και άλλους ε, λένε ε, να μην επιτρέπεται ε, αλόγιστα να διοχετεύονται πληροφορίες αλλά να λέει κανείς ότι αν ψάξει θα μπορεί να βρει νόμιμες πληροφορίες και στο επίκεντρο του όλου θέματος να τεθεί ο ασθενής και στο επίκεντρο της κοινή γνώμης. Βέβαια πρέπει κάπου να τραβήξουμε μία γραμμή μεταξύ διαφήμισης και ε, πληροφόρησης και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να βαστούμε στην αρχή εξάντε, δηλαδή πληροφόρηση η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή και να εγκριθεί προτού διατεθεί και μέσω τριών οδών των εθνικών αρχών, των αρχών και αυτών οι οποίοι θα αποδέχονται την έγκριση που μπορεί να είναι η βιομηχανία ή ο υπεύθυνο πληροφόρησης όπου δεν υπάρχει αυτό το σύστημα όπως η Σουηδία θα έλεγα ότι το σουηδικό πρότυπο είναι ένα καλό μοντέλο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η πληροφόρηση του ε, ασθενή. Δηλαδή ε, υπάρχει η ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών, exchange of good practices, ε, που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ των ασθενών είναι κρίμα λοιπόν να λέμε ότι εδώ διατυπώνουμε εξαιρέσεις. Όσον αφορά τις οδούς που διοχετεύονται οι πληροφορίες, υπάρχουν ακόμη και ιστοσελίδε. Οπότε θέλουμε ουσιαστικά <clears throat> να μην υπερβαίνουμε το όριο της πληροφόρησης και να φτάνουμε στη διαφήμιση αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η απαγόρευση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει ένας ουσιαστικός κίνδυνος και ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι ορισμένοι φοβούνται ε, και ανοίγουμε την πόρτα στη διαφήμιση εάν ε, επιτρέπουμε την πληροφόρηση στα γραπτά μέσα ενημέρωσης στον τύπο δηλαδή. Θα πρέπει γι' αυτό να επιτρέπουμε να διακινούνται πληροφορίες οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί. Ε, Καμία μέθοδος βέβαια τελικά δεν είναι τέλεια και γι' αυτό πιστεύω ότι οι τροπολογίες βελτιώνουν το αρχικό κείμενο ε, διότι περιορίζουν τη δυνατότητα ε, ε, διακινήσεως ορισμένων συγκεκριμένων ιστοσελίδων και πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διόδους τις οποίες θα επιτρέψουμε, ε, να τις παρακολουθούν, ε, να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει η ποικιλομορφία την οποία επιζητούμε και μία, ε, μία χρονιά μετά από την εφαρμογή της οδηγίας αυτής θα πρέπει να γίνει μία πρώτη αξιολόγηση. Υπάρχουν δηλαδή οι μέθοδοι για να υπάρχει η διαδικασία επιτρεπτών πληροφοριών και πρέπει να ενθαρρύνουμε να υπάρξει μια καλύτερη εξέταση του θέματος αντί να προβαίνουμε σε να απαγορεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Κράμα. Ε, πραγματικά είμαστε μέσα στην ουσία του θέματος. Ο κύριος Κράμερ δεν ξέχασε τίποτα από την περασμένη θητεία. Ε, ε, διαδίκτυο και ε, η εποχή της πληροφορικής σίγουρα θα μας κατατρέχει. Δεν πρόκειται να το αποφύγουμε. Ο κόσμος θέλει να το χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, αλλά θέλουμε να είναι και αξιόπιστη η πληροφόρηση και να ε, είναι και χρήσιμη και ωφέλιμη και όχι μόνο προπαγάνδα και διαφήμιση σκέτη. Έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως εμάς και εκεί είναι και η τέχνη, να βρούμε αυτή τη λεπτή ισορροπία. Ο Καρλ Σλούτερ. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή κύριο Φέλνερ. Επανειλημμένα έχουμε συναντηθεί, έχουμε συζητήσει για το θέμα αυτό και εμείς θέλουμε να πάμε στην διακατεύθυνση αλλά όπως λέμε συνήθως ο, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό θα χρειαστούν συμβιβαστικές προτάσεις. Εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες έχει συνταχθεί με τρόπο λανθασμένο νομίζω από την αρχή γιατί η νομοθετική πρόταση επικεντρώνεται στα δικαιώματα της βιομηχανίας, των φαρμακευτικών εταιριών και όχι στα συμφέροντα των πολιτών και στο ενδιαφέρον των πολιτών να ενημερώνονται και να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρει κανείς εκεί λύση. Στείλαμε και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας περισσότερο τα συμφέροντα των ασθενών. Εμείς θα καταψηφίσουμε η Πράσινη ε, την έκθεση αν δεν αλλάξει αυτό. Εγώ είμαι πρόθυμος να συζητήσω ό,τι θέλετε, την καλύτερη δυνατή πρόταση, αλλά πρέπει να μπει αυτό. Τώρα μπαίνουμε σε ερμηνείες, πώς θα δίδεται η πληροφόρηση, σε ποιον θα δίδεται, με ποιο τρόπο. Δεν είναι σωστή αυτή η τακτική. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, δούμε τι θα γράφει το φυλάδιο των οδηγιών του φαρμάκου που ε, συνοδεύει το φαρμακό μέσα στη συσκευασία του. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Και αρκετά χρήσιμη πληροφόρηση και αρκεί αυτή στο κάτω-κάτω. Γιατί θα πρέπει να αναγκαστούμε να εγκρίνουμε διάφορους άλλους τρόπους πληροφόρησης. Δεν μας φτάνει ε, το φυλάδιο μέσα στη συσκευασία. Η τροπολογία 83 και 119, το είπε ο Χόλγερ Κράμερ. Θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς εδώ. Τι εννοώ. Να το πω διαφορετικά προσπάθησα να το πω στην τροπολογία 83. Αλλά κάποιος που έχει οικονομικό συμφέρον να δίνει πληροφορίες για κάποιο φάρμακο, θα πρέπει να ενημερώνει, όχι να διαφημίζει. Το ίδιο λέει και η τροπολογία 172. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό. να απορριφθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση, επαναλαμβάνω. Άλλη τροπολογία για τη διαφήμιση, την τηλεοπτική. Είναι πρόβλημα. Πριν από λίγα χρόνια, θυμάστε, ε, στη δική μου χώρα είδαμε διαφημίσεις για φάρμακα ε, τα οποία δεν είναι υποχρεωτική συνταγογράφησης. Και είναι σύντομες διαφημίσεις αυτές, πολλές φορές 30 δεύτερα. Και ε, σημαντικές πληροφορίες δίνονται, τις οποίες όμως δεν μπορεί κανείς να διαβάσει, διότι δεν προλαβαίνει στη διαφήμιση. Εκτός αν έχει υψηλή ευκρίνεια μεγάλη οθόνη για να διαβάσει τα ψηλά γράμματα που προβάλλονται, εκπέμπονται με τη διαφήμιση. Οπότε δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, δεν είναι χρήσιμο. Είναι πολύ μικρό το σποτ σε διάρκεια ή είναι πολύ ασαφές. Άρα θα πρέπει απολύτως να απαγορευτεί η ειναι πολυ ασαφε διαφήμιση απολυτω να απαγορευτει η διαφήμιση γενικά για τα φάρμακα. Ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωτική συνταγογράφηση, όπω είπα προηγουμένω. Έχω και άλλη τροπολογία, την 103, που αφορά τη διαφήμιση των εμβολίων. Και πάλι δεν είναι καλό αυτό να διαφημίζονται εμβόλια. Μιλάτε για επιστημονικές μελέτες οι φαρμακευτικές εταιρείες τις δημοσιεύουν αυτές τις επιστημονικές μολέτες σαν να ήταν τίποτα αντικειμενικά στοιχεία τεκμηριωμένα και στοιχειοθετημένα. Ενώ είναι αποτελέσματα ερευνών που δεν είναι ούτε αντικειμενικά ούτε έγκυρα. Γιατί μπορεί άλλος να κάνει μια άλλη μελέτη αμέσως μετά που να αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Αν διορθωθούν λοιπόν αυτά τα κακό κείμενα ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάξει την νομοθετική της πρόταση, είμαι πρόθυμος να την υπερψηφίσω. Αλλιώ πρέπει να την αλλάξουμε εμείς την πρόταση αυτή. Και το θέμα της ενεργούς ε, αναζήτησης των πληροφοριών, της ενημέρωσης. Στη Σουηδία έχουμε ένα σύστημα που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα για την ενημέρωση των ασθενών. Πάντως καταρχήν δεν είμαι υπέρ της ιστοσελίδας και χρειάζεται έγκριση των δημοσίων αρχών γι' αυτό οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ε, ε Όσον αφορά τον Επίτροπο ο Ντάλι θα έπρεπε να αναφέρει κανείς τι είπε κατά την ακρόαση όπου λέγει ότι δεν σκοπεύω να αποσύρω την πρόταση αλλά θα την τροποποιήσω δηλαδή όταν θα έχει καταλήξει στην πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του εγώ ε, δεσμεύομαι ότι ε, θα ξανακοιτάξω το θέμα από τη σκοπιά το των πολιτών. Δηλαδή ε, θα δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο οποίο θα καταλήξει το Κοινοβούλιο και μετά θα προχωρήσει εις ε, την ε, στην αξιολόγηση και αναδιατύπωση. Η κυρία Γιανακουδάκη, ευχαριστώ για την προσπάθεια αυτή διότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια αλλά με 300 τροπολογίες προφανώς κάτι θέλει κανείς να επιτύχει. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Έχουμε πολλά προβλήματα αλλά όλοι συμφωνούμε στην πληροφορία στο δικαίωμα πληροφόρησης και στην ελευθερία πληροφόρησης και ε, ε, όπως ε, είπαμε υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή μεταξύ της πληροφόρησης και της διαφημίσεως και πρέπει να αναγνωρίζεται. Ούτε οι γιατροί είναι πολύ ευτυχείς με αυτό διότι πιστεύουν ότι η μημάθεια είναι το χειρότερο κακό και πρέπει να είμαστε καλύτερα πληροφορημένοι. Τέλος, αυτή η οδηγία ε, αποτελεί μέρος ενός πακέτου και ουσιαστικά στηρίζει και προστίθεται στις ε, δύο άλλες οδηγίες τις οποίες εξετάζουμε για την εποπτεία και την παραποίηση ε, και εξετάζουμε από διάφορες κοπιές την πληροφόρηση, όχι όμως επαρκώς, ενώ έτσι ενισχύουμε την επιτήρησή μας. Τώρα, όσον αφορά τα φυλάδια δεν νομίζω ότι επαρκούν διότι πολλοί ασθενείς τα χάνουν ή πάνε στο εξωτερικό που σας συνιστά και παίρνετε ένα φάρμακο που σας συνιστά το φαρμακείο χωρίς να καταλαβαίνετε τις οδηγίες στο πακέτο. Πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε ότι πρόκειται για διασυνοριακή προσπάθεια όλοι συνεργαζόμαστε, έχουμε διάφορες γλώσσες άρα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη αυτή η πληροφόρηση. Ε, και τώρα εδώ καταλήγω, δηλαδή δεν είναι τέλειο, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, κανείς δεν επιτυχάνει την ε, τελειότητα με την πρώτη προσπάθεια, αλλά υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, είναι σημαντική βέβαια, διότι δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να κάνει μία ελεύθερη σωστή επιλογή. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η οδηγία είναι μια καλή, ε, ένα καλό σημείο για και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια συνέχεια. Ευχαριστώ Μαρίνα. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Άννα Ρόσμπαχ, την οποία δεν βλέπω, οπότε είναι η Ντάκμα Ροντμπέρεντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Κριστό Φέλνερ προσπάθησε κάτι που είναι κάτι μεταξύ της χίλας και της χάριβδης. Δηλαδή, ουσιαστικά θεωρητικά δεν μπορεί παρά να χάσει και νομίζω ότι η προσπάθειά του επέτυχε. Διότι εδώ και 6-7 χρόνια νομίζω και περισσότερο σχεδόν από το 2001-2002 προσπαθούμε να δώσουμε πληροφορίες στους ασθενείς. Στην αρχή η Επιτροπή είχε ένα διαφορετικό πακέτο και τότε είχαμε πει στην Επιτροπή σαν Κοινοβούλιο ότι αυτό δεν επαρκεί, θέλουμε ένα μεγαλύτερο, καλύτερο πακέτο και τώρα επανέρχεται η Επιτροπή και ορισμένοι λένε δεν το θέλουμε καθόλου. Ε, μπορώ να συμφωνήσω και είμαι ευτυχής διότι τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμά στην πολιτική ομάδα δεν έχουν καταλήξει σε μια τελεσίδικη διαμορφωμένη γνώμη διότι ε, ε, ε, είναι κοινικό να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε ενημέρωση των ασθενών και αν λένε ορισμένοι ότι ε, υπάρχει ευρωπαϊκή δημοσιότης, ε, γελώ, διότι υπάρχουν, ε, υπάρχει εθνική δημοσιότητα και τρόπος με τον οποίο οι χώρες συμπεριφέρονται. Άλλη είναι η κατάσταση στη Γαλλία, άλλη στη Δανία, άλλη στη Σουηδία. Οπότε πρέπει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και να διατυπώσουμε μία σωστή πολιτική ε, ιατρική ε, για να ε, βρίσκονται σε επίπεδο ισότητος όλοι οι ασθενείς. Είμαι λοιπόν ευτυχής ή λιγότερο ευτυχής ότι ε, και είμαι πολιτικός αλλά και υπήρξα σοβαρά άρρωστη και ξέρω τι σημαίνει να μην έχω σωστή πληροφόρηση. Ε, είχα ψάξει στο διαδίκτυο πώς πρέπει ε, να θεραπεύσει κανείς την ασθένειά μου και δεν έβρισκα στοιχεία και ήμουν ευτυχής διότι είχα ένα κομπιούτερ, καταλαβαίνω αγγλικά και μπορούσα να το χειριστώ. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια ανθρώπων που δεν έχουν ε, αυτή την ευτυχία. Οπότε, ε, αν ε, δεν τους δώσουμε σωστή πληροφόρηση, θα έχουμε απαρνηθεί αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί. Εάν λοιπόν ορισμένοι μας πούν, μα θα αυξήσει το κόστος, ε, ε, γελό διότι ποιος ε, δεν θέλει ένα φάρμακο για τον καρκίνο ή ποιος πάει σε έναν γιατρό και λέει θέλω αυτό το φάρμακο παρόλο που δεν το χρειάζομαι. Αυτά είναι βλακίες. Πιστεύω ότι είναι σωστό να πούμε ε, Ζιλ, σε άκουσα πολύ προσεκτικά, αλλά έχουμε τελείως διαφορετική ε, άποψη. Ευτυχώς στην πολιτική μου ομάδα ακόμη δεν υπάρχει διαμορφωμένη γνώμη, ούτε καν να αποπέμψουμε την ε, οδηγία. Άρα το ερώτημα είναι τι θα προσφέρουμε στον ασθενή. Κανείς δεν θέλει διαφήμιση, αδιαμφισβήτησα και όλοι θα θέλαμε να κάνουμε αυτό που λέει και ο Καρλ Σλίτερ, δηλαδή πρέπει να υπάρχει διαφήμιση για τα ελεύθερα φάρμακα που μπορεί να αγοράσει ο καθένας. Αυτό δεν μας απασχολεί εδώ, υπάρχει διαφορετική νομοθεσία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και ποια είναι η ενημέρωση που χρειάζεται σε αυτό το τομέα. Όλοι συμφωνούμε, καμία διαφήμιση δεν χρειάζεται. Βεβαίω είναι επίση σαφέ ότι κάθε πληροφορία πρέπει να ελέγχεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει η βιομηχανία ούτε το θέλει ούτε πρέπει. Αλλά Παρένθεσης, η ε, βιομηχανία δεν θέλει να διαφημίσει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα διότι ο Επίτροπος Φερχόιγγεν ε, ε, δεν άφησε να περάσει κάτι τέτοιο. Επίσης και ο Κρίστο Φιέλνερ λέει πρέπει να βρούμε μια νέα λύση διότι το σύστημα που ισχύει στη Σουηδία δεν ικανοποιεί. Πρέπει να ελέγχουμε την πληροφόρηση αλλά εγώ θα ήθελα να έχουμε μία πληροφόρηση και σχετικά με την ασθένεια, όχι μόνο για το φάρμακο αλλά και για την ασθένεια. Πάρα αυτό το φάρμακο, αυτές θα είναι οι επιπτώσεις, αυτές θα είναι οι παρενέργειες, αλλά θα μπορέσει να τις μειώσεις εάν παραδείγματος χάρη κάνεις αθλήσε ή κάνεις κάτι άλλο. Δεν θα πρέπει λοιπόν επουδενή λόγο να μας σταματήσουν οι οικονομικές επιπτώσεις. Και τέλος δύο λόγια για το διαδίκτυο. Γιατί ε, ουσιαστικά πάντοτε συμφωνώ με τη συνάδελφο Λίντα Μέκερεν αλλά πάντοτε έχω πρεσβεύσει ότι υπάρχει νομοθεσία για τον λαό, όχι για την ελίτ. Η ελίτ, η εξέχουσα τάξη δεν τα χρειάζεται, μπορεί να έχει την πληροφόρηση και μπορεί να βρούνε κάποιον που θα τους πει τι ισχύει και τι όχι. Αλλά εδώ μιλάμε για το λαό που έχει γλωσσικά εμπόδια, που έχει ουσιαστικά εμπόδια και ε, αναρωτιόμαστε για την πληροφόρηση στο διαδίκτυο η οποία αποκλεί όλη την ε, γυρεότερη γενιά, τους θείους μου, τις θείες μου, τις ξαδέρφες μου όπου δεν έχουν μάθει να χειρίζονται ένα κομπιούτερ οπότε ό,τι πληροφόρηση υπάρχει πρέπει να υπάρχει και κάπου τυπωμένο να μπορεί κάποιος να το ζητήσει και να μπορέσει να το βρει είτε στο νοσοκομείο είτε στο φαρμακείο και για μένα είναι πάρα πολύ βασικό και ίσως ο συνάδελφος Κράμερ ο οποίος ε, φυγε, αναφέρθηκε εις ε, τον τύπο. Δεν θέλουμε ε, να δούμε ε, τα στοιχεία αυτά στις εφημερίδες αλλά θα ήθελα να μπορούσα τι τις πληροφορίες που μπορώ να τυπώσω από το διαδίκτυο να μπορέσω να τις πάρω και στο Σπάνταο στο Βερολίνο από το νοσοκομείο από το φαρμακοποιό. Δηλαδή, ορίστε, τι μπορώ να κάνω με αυτά τα φάρμακα και να μπορέσει κάποιος υπεύθυνο να μου δώσει στο χέρι αυτό το χαρτί να το διαβάσω. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Φέλνερ είναι στη σωστή οδό. Εγώ δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοβοηθηθούν, δηλαδή τους πιο φτωχούς, τους λιγότερο εκπαιδευμένους και για αυτούς παλεύουμε και όχι για την εξέχουσα τάξη κάποιας χώρας. Μα γι' αναζητούμε τρόπους μέσα και μεθόδους και δυνατότητες για να ενημερώνονται όλοι και για τις ασθένειές τους και για τα φάρμακά τους. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν δύο σημεία στα οποία συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Ε, όχι διαφήμιση, αλλά πληροφόρηση και η πληροφόρηση αυτή και η ενημέρωση θα πρέπει να είναι ελεγμένη. Και το θέμα είναι πώς θα φτάσει στους ασθενείς. Ποιος είναι αρμόδιος για τη διάδοση αυτής της ενημέρωσης στο διαδίκτυο ή αλλού ή και στο φυλάδιο εκείνη η σκύλα και η Χάριβδη που θα πρέπει να βρει μια διέξοδο ο κύριος Φιέλνερ για να μην χάσουμε αλλά να κερδίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Καλωσορίζω ενώπιον μας ε, μια σειρά επισκεπτών που παρακολουθούν είναι βουλευτές των Πρασίνων της Γερμανικής Βουλής στη Bundestag του Βερολίνου. Καλώς ορίσατε θερμά. Έχουμε και μια ομάδα ε, σπουδαστών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Κολονίας. Καλώς Και ακόμα και από την κάτω Αυστρία ότι έχουμε ε, της κυρίας Κάλμπαχ, ε, ομάδα επισκεπτών. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας στο Κοινοβούλιο ε, συζητάει αυτό τον καιρό το πακέτο για τα φάρμακα προς ενημέρωσή σας. Η Άνια Βάισγκέρμπερ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό ως καταναλώτρια ήδη και ως ασθενής εδώ και καιρό και θα ήθελα καταρχάς να πω ότι Είχα χαρεί ουσιαστικά που στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών που παρακολούθησα το θέμα εξ ονόματος της ομάδας μας εμφανίζεται η ίδια βασική διάκριση που βλέπουμε μόνο από ορισμένα μέλη της ομάδας και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Ροτ Μπέρεντ αυτό. Βλέπουμε και από το Γιόγκερσεν και τους ε, Πρασίνους ο κύριο Γιώργενσεν δεν είναι πράσινο, είναι σοσιαλιστή, λέει ο πρόεδρο. Σλούτερ, συγγνώμη κύριε πρόεδρε. Ε, και στην Επιτροπή λοιπόν ε, ε, εδώ δεν έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφωνία αλλά συζητούμε με μεγάλο πνεύμα συνεργασίας, επικοδομητικό και συνεννόησης και ελπίζω και οι τροπολογίες που έκανα να γίνουν δεκτές. Και εκείνοι που ζητούν απόρριψη ε, έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το θέμα επί και να το ανακαλύπτουν. Και νομίζω ότι μπορεί να στραφεί στη σωστή κατεύθυνση. Εάν επιβάλλει και η κυρία Μπέρεντ αυτό το επικοδομητικό ε, πνεύμα που δείχνει εδώ και στην ομάδα της. <laughs> Η ζωή είναι άδικη, λέει η κυρία Μπέρεντ. Ναι, ναι, το, το ξέρω. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να αγωνιστώ για τον ε, ενημερωμένο ε, ασθενή και για τον συνειδητοποιημένο ασθενή. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να φύγει η εστίαση από τη βιομηχανία, το είπε και ο Πρόεδρος, και να ε, φέρουμε στο κέντρο τον ασθενή και τον καταναλωτή. Γι' αυτό ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με τις οργανώσεις ασθενών και την άλλη εβδομάδα θα ξαναδώ πάλι μια οργάνωση ασθενών, μια ένωση ασθενών που ζητάει ξεκάθαρα νομοθεσία επιτέλους σε αυτό το τομέα, διότι όπως είπε και ο ίδιος ο σοσιαλιστής και ο εισηγητής, ε, χρειαζόμαστε ανεξάρτητη ενημέρωση και αξιόπιστη ενημέρωση. Αυτό το καιρό η πληροφόρηση υπάρχει, Dr. Google ας πούμε, στο διαδίκτυο, αλλά οι μισές πληροφορίες που δημοσιεύονται εκεί είναι μέσω θολών διάβλων όπως είπε και ο κύριος Κράμερ και είναι και ψέματα. Είναι λάθος πληροφόρηση και αυτό οδηγεί σε ανασφάλεια και παραπληροφόρηση τους ε, ασθενείς. Οπότε μην νομίζει κανείς ότι είναι όλα εντάξει και δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση. βεβαίω και χρειάζεται, διότι κυκλοφορούν και κακές πληροφορίε και λάθη στο διαδίκτυο. Και οι γιατροί το βλέπουν όλο αυτό το θέμα επικριτικά και ρώτησα εγώ πέρσι όλους τους γιατρούς που συνήντησα και μου είπαν όλοι ότι ε, θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ αν έχουμε ε, μια δικτυακή πύλη και να μπορούμε να παραπέμπουμε τους ασθενείς μας εκεί. Το θέλουμε λοιπόν αυτό. Χρειαζόμαστε ρύθμιση. Σίγουρα. Και τώρα επί της ουσίας. Βεβαίως απαγόρευση διαφήμισης, αλίμονο, αλλά έλεγχος εκ των προτέρων, όχι διαφήμιση, όχι πους να σερβίρεται διαφήμιση αζήτητη, ε, να είναι ε, ο τρόπος που είπαμε προηγουμένως, pull, δηλαδή να ε, ζητάει ο ασθενής και ο καταναλωτής την πληροφορία όταν τη χρειάζεται και όχι μόνο μέσω του διαδικτύου και με φυλάδια ενημερωτικά γιατί υπάρχουν και πολίτες πιο ηλικιωμένοι που δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι και χρειάζονται φυλάδια, όχι διαδίκτυο. Πολλές λοιπόν είναι οι δυνατότητες πληροφόρησης και όχι μόνο το διαδίκτυο. Τώρα, το φυλάδιο με τις οδηγίες στη συσκευασία του φαρμάκου, το είπαμε και στη φαρμακοεπαγρύπνηση ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είναι πολύ ευανάγνωστο αυτό. Να είναι ευανάγνωστο, να είναι γνωστές οι προφορίες και ακόμα και αχαθεί αυτό το χαρτάκι να υπάρχει δυνατότητα να το ξαναβρει κάποιο με τη μορφή αυτή την τυπωμένη. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν ηλικιωμένοι πολίτε που έχουν το φαρμακό του και χάνουν τι οδηγίε. Η κόρη του, α πούμε, δεν μπορεί ε, να βρει πουθενά τη δοσολογία γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να το ξαναβρει κάπου αλλού αυτό το φυλάδιο. Δεν δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και ε, σε πολλέ χώρε επίση δεν μπορεί να το ζητήσει ξανά ε, στο φαρμακείο. Θα πρέπει λοιπόν να δημοσιεύεται αυτό και στο διαδίκτυο. Και έρχομαι στο σημαντικότερο για μένα που είναι βασικό μου αίτημα και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ήδη το ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία όλες οι πολιτικές ομάδες το υποστήριξαν αυτό που ζήτησα. Και τι είναι αυτό. Ε, ε, πέρα από τα φυλάδια και την πολύ σημαντική ενημέρωση στα διάφορα κράτη-μέλη να υπάρχουν ιστοσελίδες βάσει του σουηδικού παραδείγματος. Στη Σουηδία είναι καλό το σύστημα ε, με ελεγμένη ενημέρωση, ε, ε, μια δικτυακή πύλη που χρησιμοποιούν 4 εκατομμύρια πολίτες και θυμίζω ότι η Σουηδία έχει 8 εκατομμύρια κατοίκους. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και είναι ευέλτιστη πρακτική, μπορούν να την υιοθετήσουν και τα κράτη-μέλη και να δημιουργήσουν τέτοιες ιστοσελίδε. Και συμφωνώ με την κυρία Ροτ Πέρεντ, να μην είναι αφετηρία το φάρμακο, αλλά ε, η ασθένεια. Δηλαδή, αν έχω υπέρταση, να με ενημερώνουν και για το σωστό τρόπο ζωής, τη σωστή ε, διατροφή, την άθληση. Όχι μόνο πάρει το τάδε φάρμακο να σου πέσει πίεση. Να έχουμε πληροφόρηση και για ε, την ασθένεια και με τρόπο που να βοηθάμε τον ασθενή. Αυτά. Μου είπε ο εισηγητή ότι είναι πρόθυμο να συζητήσει και την ιδέα αυτή. Ελπίζω να περάσουν οι τροπολογίε μα και αν συμφωνήσουν και άλλε πολιτικέ ομάδε με την 100 και την 112. Παρακαλώ, ξανακοιτάξτε τη και την 74 για την αιτιολογική σκέψη. Να τα δούμε όλα αυτά παράλληλα πάντα με τα φυλάδια μέσα στη συσκευασία του φαρμάκου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάισκερπερ. Ο Χόρστ Σνέλχαρτ, επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν πιστεύω ότι ο εισηγητής ε, ε, μας οδηγεί στο να χάσουμε αλλά κερδίσαμε πολλά στη συζήτηση διότι θυμάμαι την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπήρχε αυτό που δημιουργεί την αντίδραση σε ορισμένες πλευρές του Κοινοβουλίου και με την αντίδραση αυτή οδηγήσαμε, ε, οδηγηθήκαμε στο σημείο εδώ που λέμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο ζητάμε πληροφόρηση και όχι διαφήμιση όλα αυτά είναι σαφή Βέβαια το ερώτημα είναι πού είναι το όριο και ποτέ δεν μπορούμε να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή τόσο σαφώς και να λέμε ότι πληροφορούμε χωρίς καθόλου να διαφημίζουμε. Μετά από πέντε χρόνια πιστεύω ότι όταν θα κάνουμε μια επαλήθευση θα δούμε ότι δεν έχουμε επιτύχει 100% διότι πάντοτε ε, ε, θέλουμε να μην υπάρχει και τόση γραφειοκρατία, είναι κάτι που μας απασχολεί ε, και νομίζω ότι εδώ μετά από πέντε χρόνια πρέπει να υπάρξει μία επαλήθευση, να δούμε τι διεξήχθη και εάν ο ασθενής όντως έχει την ενημέρωση την οποία απαιτεί. Άκουσα όμως τους συναδέλφους οι οποίοι είπαν ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει και στο διαδίκτυο αλλά αν δεν υπάρχει κομπιούτερ τι θα κάνουμε. Ε, εφόσον υπάρχουν συνεχώς καινούργιες πληροφορίες ε, δεν μπορούμε εμείς να του τα δώσουμε όλα στο πιάτο. Θα πρέπει και ο ασθενής να φροντίσει ό,τι πληροφόρηση λαμβάνει να την διατηρεί. Και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η πρόταση αυτή να επιτρέπει στη συσκευασία να υπάρχει ε, μία συνοπτική ενημέρωση κατά τρόπον ώστε ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το φάρμακο να μπορέσει να ενημερωθεί. Βεβαίως ε, ε, με άλλες, άλλους τρόπους θα μπορέσει να μάθει και ποιες άλλες θεραπευτικές δυνατότητες υπάρχουν έχει καλώς αλλά δεν χρειάζεται ο, ο κατασκευαστής του φαρμάκου να γράψει επάνω ότι μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα με αυτό το, φά, το φάρμακο ή μπορείς για αυτή την ασθένεια να χρησιμοποιήσεις άλλα φάρμακα. Δεν πρέπει να ζητάμε πάρα πολλά. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Και Γι' αυτό θα κάνουμε αυτή την πρόταση, θα την παρακολουθήσουμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. θεωρώ ότι έκανε σωστή εργασία ο, ο και τον ευχαριστώ. Λοιπόν, η αισιοδοξία του Χόρστ Σνέλχαρτ, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ο Πέτερ Λίζε όμως τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή, ε, τον Κρίστοφερ Φέλνερ, διότι πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο δεν επέτυχε η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, να διαχωρίσουμε σαφώς την πληροφόρηση από τη διαφήμιση και αυτό πρέπει να επιτευχθεί καλύτερα από ό,τι το επιτυγχάνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η τελική λύση κατεμένα είναι κάτι ανάμεσα στην πρόταση του Κρίστοφερ Φέρνελ και του ε, κυρίου Βερνιό. Ε, νομίζω ότι ε, δεν μπορούμε να αποπέμψουμε την πρόταση αυτή διότι θα μας κοστίσει χρόνο ο οποίος δεν μας περισσεύει και θέλουμε ε, να ενισχύσουμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου το οποίο έχουμε διαπραγματευτεί σκληρά με τον κύριο Μπαρόζο. Άρα θα πρέπει το κοινοβούλιο όπως φροντίζουμε να διατυπώσει μία πρόταση η οποία θα είναι η βάση συζητήσεως. Τρία θέματα όμως ε, μου είναι ουσιαστικά εάν διατηρήσουμε την πρόταση αυτή. Ήδη υπάρχει καλή και ανεξάρτητη πληροφόρηση στο διαδίκτυο και πολλές φορές θυμώνω διότι ο κύριος Φερχόγγεν σαν γερμανικός σαν γερμανός επίτροπος λέγει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι νέο αλλά στη Γερμανία υπάρχει το Ινστιτούτο για την ποιότητα των φαρμάτων που είναι πολύ αντικειμενικός οργανισμός και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη δικιά του πορεία. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένα φάρμακα σε ορισμένες χώρες όπου θα άξιζε η προσπάθεια των κρατών μερών ε, ε, ε, και των, βιομηχανιών να υπάρξουν οι οδηγίες χρήσεως όχι μόνο στις μεγάλες γλώσσες αλλά και σε μικρότερες, στις ουγγαρές, ή ε, ε, σε κάποια άλλη μικρή γλώσσα. Ε, επίσης δεν υπάρχει λόγος ε, η αποδεκτή ε, πληροφόρηση να υπάρχει σε όλες τις ε, δυνατές γλώσσες. Δηλαδή στη Γαλλία θα πάρετε οδηγίες χρήσεως που να είναι γαλλικά και ενδεχομένως γερμανικά. Αλλά θέλετε, επανέρχομαι πάλι στα ουγγαρέζικα, γιατί να μην μπορεί να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο διαδίκτυο για γιατί να μην βελτιώσουμε τη συσκευασία ε, κατά τρόπον ώστε να είναι πιο ευανάγνωστες οι οδηγίες χρήσεως διότι εκεί θα έχουμε τις ουσιαστικές πληροφορίες θα μου πείτε είναι δύσκολο όλα είναι βασικά αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά αυτό προποθέτει ότι ο ασθενής καταλαβαίνει τα πάντα αλλά εγώ σαν γιατρός έχω μια εμπειρία που λέει ότι ο ασθενής δεν διαβάζει καν τις οδηγίες χρήσεως δεν διαβάζει καν τις προειδοποιήσεις ε, για τις παρενέργειες και ούτε καν ότι ε, το φάρμακο πρέπει να παίρνεται υπό ορισμένε συνθήκε όπως τους έχει συνταγογράψει ο, ο ιατρός αλλά ποτέ δεν είδα έναν ασθενή ο οποίος είπε δεν πήρα το φάρμακο γιατί ε, ε, δεν ε, ξέρω ποιες είναι οι παρενέργειες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κουτάκι όπου όλα να αναφέρονται σαφώς. Επίσης ελέγχθη ότι αυτός ο οποίος θα λαμβάνει την άδεια δεν είναι υποχρεωτικά η βιομηχανία. Αλλά αυτό είναι θεωρία, διότι ουσιαστικά όποιος έχει την άδεια να κυκλοφορήσει ένα φάρμακο είναι επιχειρηματίας και πρέπει να προσέξει, διότι τι ε, συμφέρον έχει η φαρμακευτική επιχείρηση ε, για ε, να πουλήσει ένα φάρμακο ή να το δώσει προς διάθεση και σε άλλους εάν δεν βελτιώσει τις πωλήσει του. Άρα θα πρέπει να υπάρξει καταρχήν μία άδεια για να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια και συμφωνώ με τον κύριο Χατζημαρκάκη, την κυρία Βάις Γκέρμπερ, ότι το σύστημα ίσως λειτουργεί ε, σωστά στην ε, Σουηδία χωρίς να χρειάζεται προκαταρκτική αδειοδότηση και αυτό να αποτελέσει μία εξαίρεση. Αλλά για τα υπόλοιπα κράτη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να εξετάσουμε την ε, χορήγηση αδείας προτού κυκλοφορήσουν οι πληροφορίες διότι εγώ δεν είμαι μεν νομικός αλλά αν επί ε, επιτραπεί να ελέγξουμε τις οδηγίες χρήσεως το τι γράφεται πάνω γιατί δεν είναι δυνατόν οι επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες δεν δίνουμε τώρα να μην διατίθενται επίσης εφόσον έχουν ελεγχθεί εκ προημίου δηλαδή ε, όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν ε, εγκριθεί από κάποια αρχή να μπορούν να διατεθούν. Η νομική υπηρεσία πρέπει να μας πει πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι ό,τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια αυτά μπορεί να διατεθεί ε, με διάφορους τρόπους που δεν ήταν διαθέσιμοι μέχρι τώρα και φτάνω στο πρώτο τελευταίο σημείο μου. Δηλαδή συμφωνώ με αυτό που είπε η Ντάκμα Ροντμπέρεντ. Χρειαζόμαστε ένα έντυπο υλικό. Δηλαδή ε, ε, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο φυλάδιο διότι μπορούμε ε, να προστρέξουμε στο διαδίκτυο και υπάρχει μία ενημέρωση η οποία σε ορισμένα σημεία είναι συγκρίσιμη με την εφημερίδα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι μπορεί κανείς να δημοσιεύσει κάτι στο Google ή στο διαδίκτυο γενικό ε, που δεν επιτρέπεται να δημοσιευτούν σε μία εφημερίδα. Πρέπει να ε, ε, διαχωρίσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Και τέλος ένα πολύ βασικό θέμα είναι ότι δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι ε, ε, δεν διαθέτουμε αναγκαία φάρμακα ή στους ασθενείς. Ε, θα πρέπει να τους πούμε ότι υπάρχει μία δυνατότητα την οποία ίσως δεν είχαν σκεφτεί και υπάρχουν και οργανώσεις ασθενών που είναι πιο καλά πληροφορημένες ε, από ότι ε, οι ιατροί. Αλλά η λανθασμένη πληροφόρηση μπορεί να ανεβάσει το κόστος και μπορεί να οδηγήσει σε παρενέργειες. Διότι αν δεν γίνει σωστή οριοθέτηση, συμφωνούμε ότι θέλουμε να το οριοθετήσουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο ε, παρισφρήσει διαφήμιση ή κάτι που λειτουργεί σαν διαφήμιση σαν μονοπλευρή ενημέρωση τότε τα ε, φάρμακα τα οποία προωθούνται είναι τα καινοτόματα τα οποία είναι και τα πιο ε, ακριβά και που έχουν πολλές παρενέργειες. Δηλαδή χρειάζεται η φαρμακοεποπτεία. Αυτή χρειάζεται διότι πρέπει να διαπιστώσουμε μετά την αδειοδότηση εάν παρουσιαστούν παρενέργειες οι οποίες προηγουμένως δεν γνωρίζαμε. Εάν λοιπόν ε, επιτρέψουμε ε, να ισχύσει στην αγορά ένας μηχανισμός που θα τα προωθεί περισσότερα θα έχουμε ε, μεγαλύτερο κόστος και ίσως περισσότερες παρενέργειες. Άρα πρέπει να υπάρχει καλή ποιοτική ε, ενημέρωση, να αποκλείσουμε τη διαφήμιση και όπως είπε ο Κρίστοφερ Φέρνερ θέλουμε χρόνο. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον Ιούνιο, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να τα εξετάσουμε. Ευχαριστώ Πέτερ Λίζε. Και τώρα καταναλώσαμε περισσότερο χρόνο από είχα υπολογίσει θα έρθει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου σε λίγο και είναι και πάντα στην ώρα του. Άλλους ε, δύο να ακούσουμε, δύο, δύο καθένας για να προκάνουμε. Δύο λεπτά ο καθένας. Ο Γιάννος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Δύο λεπτά τι να πω. Ε, θα επικεντρωθώ σε μία και μόνη τροπολογία. Ο κύριος Σλούτερ μπορεί να πιστεί ε, νομίζω, γιατί μία από τις τροπολογίες αυτές είναι περιττή. Ο κύριος Σλούτερ είπε να μην γίνεται τηλεοπτική διαφήμιση για φάρμακα, φάρμακα που δεν απαιτούν ε, ιατρική συνταγή όχι, εντάξει, να απαγορευτούν οι διαφημίσεις, αλλά αυτή τη στιγμή ο κανονισμός που ισχύει ορίζει ότι φάρμακα που δεν χρειάζονται συνταγή επιτρέπεται να διαφημίζονται στη τηλεόραση. Εφόσον λοιπόν αυτό επιτρέπεται, διαφημίζεται το προϊόν αυτό, το φάρμακο και το αγοράζουν περισσότερο οι ασθενείς. θα πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους ασθενείς. Εξάλλου αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούρια. Τα τελευταία 20 χρόνια ισχύει η διαφήμιση και δεν αποδείχθηκε πουθενά ότι σε φάρμακα που δεν θέλουν συνταχή ε, αυξήθηκε η χρήση τους λόγω της τηλεοπτικής διαφήμισης. Δεν έχει ε, αυτό αποδειχθεί γιατί και από τη τηλεόραση να απαγορευτεί μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει διαφήμιση ε, στο ραδιόφωνο ή στις εφημερίδες με τις ίδιες προφορίες. Στη συνέχεια, είναι σαφείς οι κανόνες για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και καλά ρυθμισμένα αυτά, ιδιαίτερα ε, ως προς το περιεχόμενο της διαφήμισης για το φάρμακο. Εάν το απαγορεύσουμε αυτό τώρα στην τηλεόραση, τότε ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταφεύγουν ε, γιατρούς για να παίρνουν φάρμακα υποχρεωτικής συνταγογράφησης. Έτσι και να ε, θα αυξηθεί επομένως ε, και το κόστος της υγείας γιατί θα πληρώνουν και την επίσκεψη. Κυρία Μακάβαν. Um, Νομίζω ότι ε, αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση που είπαν πολλοί, δηλαδή για τις πληροφορίες για τον ασθενή, να μιλήσουμε για δημόσια υγεία και για τον ασθενή πρωτίστως, δεν θα δω τις ε, φαρμακοβιομηχανίες, τότε μόνο θα έχουμε τη σωστή απάντηση. Πολλοί είπαν ότι ίσως πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση. Κανένας όμως δεν αρνήθηκε πληροφορίες προς τον ασθενή. Το ζήτημα είναι πώς θα διοργανωθούν ε, πρόσφατα ένας φίλος ε, διαγνώστηκε, μία φίλη διαγνώστηκε με μία χρόνια ασθένεια και της είπα τι θα επιθυμούσε. Είπε ότι θα ήθελα να βρεθώ σε ένα ουδέτερο δαφός και να μου πούν τι μπορώ να κάνω για την κατάστασή μου, τι είναι διαθέσιμο στην αγορά, τι ξέρουμε για αυτή την ασθένεια και τι επιλογές έχω δεν θέλουν να πάνε στην ιστοσελίδα μιας ε, φαρμακοβιομηχανίας για να δούνε ποια είναι τα υπέρ και τα κατά ενός φαρμακού. Έχω ασχοληθεί με το θέμα της ε, φαρμακογρύπνησης και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή να αποστείλει ένα σημείωμα προς όλους, να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει από τον οργανισμό του Λονδίνου γιατί ήδη είναι διαθέσιμες πολλές πληροφορίες. Μετά θα δούμε τι προτείνεται στην νομοθεσία μας περί φαρμακοεπαγρύπνησης, γιατί εκεί έχουμε όλα τα φάρμακα, όλες τις πληροφορίες στην ευρωπαϊκή δηλαδή πύλη και στη συνέχεια κάθε φαρμακοβιομηχανία να έχει τη δική της ιστοσελίδα. Συμφωνώ με την Dagmar ότι δεν αρκούν οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα. Δηλαδή, θα πρέπει κανείς να μπορεί να γράψει στις εθνικές αρχές, να λάβει τις πληροφορίες από τις εταιρείες. Αλλά νομίζω ότι επειδή τα περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα, θα μπορούσε να μας δώσει μία ανακοίνωση η Επίτροπη. Θα ήθελα να πω στον κύριο Φέλνερ ότι γνωρίζουμε το ιστορικό της πρότασης, αλλά θα πρέπει εσείς και οι σκιώδεις να προβάλλετε τροπολογίες έτσι ώστε να δίνετε πληροφορίες προς τον ασθενή και μόνο έτσι θα τύχετε υποστήριξης. Δεν μας ενδιαφέρει τι μπορούν να ε, βάλουν οι φαρμακοβιομηχανίες, τι διαφημίσεις μπορούν να εισαγάγουν, πού και γιατί. Τα κράτη-μέλη θα μας δώσουν πληροφορίες στα εθνικά, στις εθνικές ιστοσελίδες. Ανδρές Περέλ. Ευχαριστώ. Εντάχει, διότι όλα ελέγχθησαν. Δέχομαι τις προθέσεις του εισηγητή. Θέλουμε να περισσώσουμε το κείμενο, αλλά συμφωνώ με τον κύριο Πανιό Δηλαδή το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε είναι να αποσύρουμε αυτή την ε, πρόταση. Δεν είναι καλή ή κακή επειδή έχει πολλές ή λίγες ε, τροπολογίες. Οι τροπολογίες όμως πρέπει να βελτιώνουν το κείμενο, αλλά εδώ κανένας δεν ήταν σε θέση να πει ότι είναι καλή η οδηγία, γιατί είναι αδύνατο να πούμε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό το κείμενο θα πρέπει να το αλλάξουμε άρδιν. Το πρόβλημα είναι ότι το μόνο που σώζουν, περισσώζουμε είναι ο τίτλος, δηλαδή πληροφορίες προς τον ασθενή. Όμως ε, δεν είναι συνεκτικό το κείμενο. Δεν μιλάμε για άρνηση πληροφόρησης. Εγώ θέλω πληροφόρηση προς τον ασθενή, αλλά μιλάμε για προϊόντα τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν μετά από, ή να δοθούν μετά από συνταγογράφηση. Δεν πρόκειται για ένα CD ή για μια οικιακή συσκευή. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος δίνει τις πληροφορίες και πώς τις δίνει. Και δεν μας το διασαφηνίζει αυτή η οδηγία. Δεν υπάρχει όριο μεταξύ πληροφορίας και διαφήμισης. Θα πρέπει να κατανομάζουμε τα πράγματα όπως έχουν. Μπορούμε και με τις τροπολογίες να πούμε στην Κομισιόν ότι το κείμενο δεν είναι σύνεπες. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν στο Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλους έξι μήνες. Δεν θα πρέπει να είμαστε στην πλευρά των φαρμακευτικών βιομηχανιών και όχι στην πλευρά των ασθενών. Ευχαριστώ. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή συζήτηση και ο εισηγητής ε, πρέπει να δώσει τις τελευταίες πινελιές εφόσον αυτός θα πρέπει να καταλήξει στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πρόθεσή μου ήταν να μην μιλήσω για θέματα αρχής γιατί είναι κάτι που το θεωρώ δεδομένο. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνουμε ότι τασόμαστε κατά της ε, διαφήμισης. Το έχω πει τόσες μα τόσες φορές αυτό και όλοι συμφωνούν. Κανένας μας δεν θέλει διαφήμιση. Δεν έχει νόημα να το επαναλαμβάνω ad Έχω όμως την εντύπωση, με βάση αυτά που είπε και ο τελευταίος ομιλητής, ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό το είπε και ο σκιώδης των σοσιαλιστών. Το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά της πρότασης, αλλά να, δούμε τις, να πάρουμε τις καλές ιδέες. Ο κύριος Μπαρνιό έφτασε σε πολύ καλές ιδέες, οι οποίες δεν συζητήθηκαν. Δεν θα ήθελα να αρχίζουμε εκ του μηδενός κάθε φορά, να μιλάμε για το περιεχόμενο, γιατί θα βρεθούμε στην ίδια θέση και χάνουμε χρόνο, όπως χάσαμε από το 2001. Εγώ θέλω να εργαστούμε. και ελπίζω αυτό να ισχύει και για σας. Το μόνο θέμα το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο σήμερα αφορά τις δαπάνες στον τομέα υγείας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σαφείς. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ενημερώνονται ή δεν πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες για τη συμπίεση του κόστους. Υπάρχουν πάντα πολύ καλοί λόγοι γιατί πρέπει να περιορίσουμε τη διαφήμιση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σταματάμε τη διαφήμιση για να συμπιέσουμε το κόστος. Ο κύριος ε, Κάρμερ αναφέρθηκε σε ορισμένα σημεία τα οποία με απασχόλησαν. Πιστοποίηση των ιστοσελίδων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαδικτυακές πύλες που δεν ανήκουν στις φαρμακοβιομηχανίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πιστοποίηση από, κάποιον τομέα, από κάποιο φορέα της αγοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης. Διακόπτει ο Πρόεδρος θα πρέπει να περιοριστείτε γιατί περιμένουμε τον ε, προσκεκλημένο μας. Ε, θα ήθελα να πω δύο πράγματα εν τέλει. Ούτε ένα λεπτό δεν χρειάζομαι. Πιστεύω ο... και θα πρέπει να πω στον κύριο Σλούτερ ότι η οδηγία όπως είχε όταν την πρωτολάβαμε, τασόταν άρδιν υπέρ της βιομηχανίας και όχι υπέρ των ασθενών. Αυτό το καταφέραμε με 300 τροπολογίες και θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Να ακούμε οι μεν τους δε. Από αυτή τη συζήτηση συμφωνήσαμε σε πολλά. Ε, όταν ε, μιλήσαν ο Καρλ και η Άνια Βάισκερμπερ, είδα ότι συμφώνησαν. Και αυτό είναι ένα πολύ σωστό μήνυμα. Εάν δεν ε, υπάρχουν ε, συμπαγείς αντιρρήσεις, νομίζω ότι θα φτάσουμε σε λογικούς συμβιβασμούς, έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν καλύτερες πληροφορίες. Ας σταθούμε σε αυτό και ας αρκεστούμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Είναι μια πολύ σημαντική ε, έκθεση για αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι σωστά ενημερωμένοι και ελπίζω ότι θα υπάρξει ευρεία συνένεση στην Επιτροπή που θα βοηθήσει αυτή την έκθεση και ε, θέλω να ε, να καλωσορίσω τους ε, ε, επισκέψεις της Κάριν Κάλενμπαχ που ήρθε στην Επιτροπή μας και επειδή ο πρόεδρος βρίσκεται πρώτων θυρών και θα έρχεται να μας επισκεφθεί ε, πρέπει να του επιτρέψουμε να εισέλθει. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρό μας, τον ε, κύριο ε, Μπούζεκ. Σας καλωσορίζω στην ε, Επιτροπή μας, η οποία είναι η μεγαλύτερη Επιτροπή που επιτελεί νομοθετικό έργο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Τώρα μιλήσαμε για το πακέτο των φαρμακευτικών σκευασμάτων, πληροφορίες προς τον ασθενή, προς τους ασθενείς, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά μας απασχολούν και άλλα θέματα όπως οι κλιματικές αλλαγές. Και χαίρομαι διότι ε, θα μας μιλήσετε για τα αποτελέσματα της επίσκεψής σας ε, στην Κίνα. Και εγώ βρέθηκα στην ίδια πόλη, αλλά δεν σας είδα, είναι τεραστίων διαστάσεων η πόλη. Είχαμε πολλές επαφές με αυτή τη νέα αναδυόμενη ε, δύναμη στη Παγκόσμια Σκακέρα και συμμετείχα και με τον Ζακ Ντελόρ σε ένα γεγονός στα πλαίσια μιας μελέτης για τη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ενέργεια. Ξέρουμε ότι η ενέργεια ε, ασχολείται και με τον ε, εφοδιασμό προμηθειών και με μεγάλη μου χαρά θα σας δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις ε, δικές σας ιδέες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Κατά την προηγούμενη θητεία, για πέντε χρόνια, συμμετείχα στην Επιτροπή Ένδη Ξέρετε τα τέσσερα βασικά σημεία που θα σας παρουσιάσω. Πρώτα μιλάμε για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια, ε, την, τον εφοδιασμό των ε, προμηθειών, ενεργειακών προμηθειών, αλλά θα ήθελα να αρχίσω από τα πιο γνωστά θέματα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών Και θα πρέπει να ζητήσουμε από τις μεγάλες επιχειρήσεις ενεργειακής προμήθειας, προμήθειας ποιες είναι οι επενδύσεις μακροχρόνια για την ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας και για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις οι επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική επί του θέματος. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία για το τέταρτο σημείο που θα σας ε, θίξω. Οι προσδοκίες του πολίτη θα πρέπει να υπάρχει ε, συμπίεση του κόστους ενέργειας, διότι αυτό είναι πολύ καλό και για τους πολίτες και για την ανταγωνιστικότητα της αγοράς μας. Δεν ξέρουμε πού θα κινηθούν αυτές οι ταπάνες, αλλά θα πρέπει να είναι χαμηλές. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια κοινή προσέγγιση επί του θέματος, διότι θα είμαστε πιο επιτυχείς εάν έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Και μας ενδιαφέρει και η ε, ενιαία αγορά βεβαίως. Έχουμε προετοιμάσει μία νομοθεσία πρόσφατα, τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια, το δεύτερο και το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Όλα τα πακέτα για τα κλιματικά ζητήματα, ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα ζητήματα. Επίσης και η ανταλλαγή ε, αερίων θερμοκηπίου. Όπως ξέρετε θα γίνουν διαβουλεύσεις για την νέα ενεργειακή αποδοτικότητα εν ώψη του 2020 Υπάρχουν πολλά συστήματα επιτάπητος, πολλά ε, θέματα βρίσκονται στη διαδικασία ε, προετοιμασίας και βεβαίως και η ρύθμιση για την προμήθεια ε, φυσικού αερίου, η οποία γνωμοδο... επί της οποίας γνωμοδότησε η Ήτρε και θα ψηφιστεί τον Ιούλιο από την Ολομέλεια. Και έχουμε και άλλα παλαιότερα ζητήματα, την ενίσχυση της συνεργασίας η προμήθεια ενέργειας από τους εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφοροποίηση, αποδοτικότητα της ενέργειας, η χρήση της και οι πιθανές διασυνδέσεις. Υπάρχει κάποια πρόταση, υπάρχει πρόταση για να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε πολιτικά την όλη πρωτοβουλία να ενδυναμώσουμε αυτή την πρόταση. Και τέσσερα είναι τα βασικά σημεία. Η εφαρμογή, καταρχήν, όλων των κανονισμών που προαποφασίστηκαν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια. Δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Έχουμε το δεύτερο ενεργειακό πακέτο και το τρίτο που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Και ορισμένα άλλα για τα ανανεώσιμα, το CCS. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο ε, αντιτιθέμεθα σε ορισμένους ε, κανονισμούς, πώς μπορούμε να τους βελτιώσουμε, να τους ενισχύσουμε. Το δεύτερο θέμα είναι η ενίσχυση συνεργασίας σε σχέση με τα ενεργειακά δίκτυα. Εάν θέλουμε δηλαδή να συμπληρώσουμε την ενιαία αγορά, θα πρέπει να δούμε τα ενεργειακά δίκτυα, πώς μπορούμε να τα ενισχύσουμε. Δεν υπάρχουν επαρκή δίκτυα, δηλαδή διασυνοριακές διασύνδεσεις. Τρίτον, κοινά ταμεία για τη χρηματοδότηση των νέων ενεργειών. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα ενεργειακής επάρκειας για την προστασία του κλίματος. Μιλάμε για βιομάζα, ηλιακή, αιωλική και ούτω καθεξής. Αλλά δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Αυτό αφορά και την ε, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και τα πυρηνικά μέσα στα πλαίσια της Ευρατό. Και το τέταρτο σημείο που αφορά την απαρχή της συνεργασίας θα πρέπει να δούμε πώς έχουν οι κοινοπραξίες παροχής φυσικού αερίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μεγάλες εντάσεις βεβαίως ως προς τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές μεταξύ κρατών μελών. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Θα, θα προτιμούσαμε να υπάρχει συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προμήθεια ενέργειας. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και βεβαίως ποια είναι η θέση των μεγάλων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ για να τους δώσουμε κίνητρα για έρευνα, για ε, καινοτομία. Σε σχέση με αυτά που είπε ο πρόεδρος στην αρχή, επισκεφτικά της είπα, είναι ζωτική σημασία συνεργασία μας και με τις είπα, αλλά θα ήθελα να σας πληροφορήσω για τις συναντήσεις μου στην Κίνα ήρθα σε επαφή με τον επικεφαλής του Κοινοβουλίου, τον Πρωθυπουργό, δύο υπουργούς, τον Υπουργό Ενέργειας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ως προς τις κλιματικές αλλαγές καταρχήν, πολλά ελέγχθησαν κατά τις διαπραγματεύσεις, μπήκαμε σε λεπτομέρειες, Έχω όλα τα στοιχεία διαθέσιμα, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από τη δική τους πλευρά. Ο Υπουργός ο υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις φαίνεται να είναι υποστηρικτικός. Όταν μίλησα με τον Υπουργό Ενέργειας ε, απεκόμισα το ακριβώς αντίθετο. Δεν δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Τον ενδιαφέρει η ανάπτυξη της Κίνας στον τομέα της ενέργειας δεν ενδιαφέρεται τόσο για κλιματικά ζητήματα, άρα ίσως να υπάρχει και μία ενδοκυβερνητική ε, διαφωνία. Θέλουν να υποστηρίξουν τις ανανεώσιμες, αλλά όχι λόγω κλίματος, αλλά λόγω ασφάλειας εφοδιασμού. Δεν θέλουν να εξαρτώνται, να είναι εξαρτώμενοι. Αυτό καθίσταται σαφές. Άρα ανανεώσιμες για αυτούς σημαίνει μεγαλύτερη ε, εφοδιαστική επάρκεια και ασφάλεια. Αυτό αφορά και την ε, απόδοση, την αποδοτικότητα. Θέλουν τη συνεργασία. Είναι ένας ε, τομέας τον οποίο εγώ τους έκανα να ανακαλύψουν. Άρα για μας διανοίγεται μία νέα δυνατότητα δηλαδή να προβάλλουμε τις δικές μας τεχνολογίες. Ως προς τον άνθρακα, χρησιμοποιούν 80% άνθρακα για την ηλεκτροπαραγωγή και δεν θέλουν να αλλάξουν τις ε, αναλογίες τα ποσοστά. Δηλαδή, σε 10 χρόνια πάλι θα είναι 80% της ηλεκτρικής ε, παραγωγής που θα εξαρτάται από τον άνθρακα και 20% ανανεώσιμες. Ίσως και πυρηνικά ημέρη. μέρη. Αλλά η ζήτηση ηλεκτροπαραγωγής θα είναι διπλάσια από τη σημερινή. Αν θέλουν λοιπόν να κρατήσουν τις ε, αναλογίες αυτές, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να διπλασιάσουν τις ανανεώσιμες και προσπαθούν να το κάνουν αυτό, αλλά όχι για να αλλάξουν την ποσοστιαία αναλογία, αλλά για να την κρατήσουν. Γιατί η ζήτηση σε παροχή ηλεκτρισμού και ενέργειας θα αναπτυχθεί άρδιν στην Κίνα. Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Η ανάπτυξη ανανεώσιμων σημαίνει ότι κρατάμε τις ίδιες αναλογίες. 70 με 80% ηλεκτρισμού που θα παράγεται από άνθρακα. Και τώρα έχουν μία πρόταση δική τους για το πρόγραμμά τους. Τρία δις τόνους ετησίως. Τρία τόνους ετησίως ε, παραγωγή άνθρακα. Δεν τους ενδιαφέρει η αποθήκευση του άνθρακα. Και γι' αυτό το ζήτημα για μας είναι ζωτικής ε, σημασίας και για σας, την Επιτροπή Έμβη, που ηγείστε αυτού του ζήτηματος. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους ε, Κινέζους με την παραγωγή άνθρακα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ε, άνθρακα. Άρα τι θα γίνει σε σχέση με την ίχνη λάτηση και ε, αποθήκευση του άνθρακα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ε, ελέγξει. Μιλάμε για 12 εγκαταστάσεις ως προς το CCS. Και για να δώσουμε αυτή την τεχνολογία στους Κινέζους σε 5, 10, 15 χρόνια, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτή, να την έχουμε αναπτύξει. Πρέπει να προβλέψουμε το μέλλον. Θέλουμε να σταματήσουν την παραγωγή άνθρακα και τον ηλεκτρισμό από τον άνθρακα. Δηλαδή το 35% ίσως γίνει 50%, ίσως γίνει 60%, ίσως είναι καλύτερα από πλευράς εκπομπών, αλλά οι εκπομπές θα υπάρχουν. Τι θα γίνει με τη συνεργασία ως προς τα πυρηνικά. Θέλουν να προβούν στην εγκατάσταση νέων σταθμών, αλλά ως προς τον άνθρακα δημιουργούνται ε, όλο ένα και μεγαλύτερες και περισσότερες μονάδες παραγωγής άνθρακα πρέπει να ξέρουμε τι επακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι ανοιχτή προς τη συνεργασία, πνευματικά δικαιώματα. Μας δώσανε θετική απάντηση, αλλά δεν ξέρω πώς θα αξιολογηθεί στο μέλλον. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα είχα να σας πω, αλλά θα σταματήσω εδώ για να μου υποβάλλετε και ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για όλες αυτές τις ε, πληροφορίες για την Κίνα και την παρουσίαση ορισμένων ιδεών. Συνεργαζόμαστε στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε και το ιστορικό αυτό συνεργασίας. Είχαμε την ΕΚΑΧ, στη συνέχεια την ΕΒΡΑΤΟΜ και εδώ και πολλά χρόνια οι ανανεώσιμες αποζητούν μία συνθήκη. Μετά από 50 χρόνια υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει σε αυτό το τομέα και έχουμε και έναν επίτροπο ενέργειας κάποιον από τη χώρα μου, ο οποίος έχει δεσμευθεί και ε, επισκέπτεται τον κόσμο για να αναζητήσει απαντήσεις όπως και εσείς η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Νιγηρία και άλλες χώρες, για αυτές τις χώρες ε, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να βρούμε μία λύση για τον άνθρακα. Γιατί ο άνθρακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και το θέμα του CCS της αποθήκευσης του άνθρακα είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα είναι πώς ε, αυτή η τεχνολογία φτάνει στην Κίνα, πώς θα φτάσει στην Κίνα. Υπάρχουν και οι μηχανισμοί καθαρής ενέργειας, η μεταφορά τεχνολογίας, όλα αυτά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Δεν μπορούμε να τα χειριστούμε ε, ομαδών βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Υπάρχει πληθώρα ερωτήσεων. Ε, Ρίτσαρντ Ζέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω τον Πρόεδρο Μπούζεκ και να το πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι ε, μπορεί να μοιραστεί τις εμπειρίες του μαζί μας. Ε, τα ε, θέματα που έθεσε είναι πολύ επίκαιρα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι αν συζητάμε τα θέματα αυτά σαν νομοθέτες πρέπει καταρχήν να εξετάσουμε αν χρειαζόμαστε νέες ρυθμίσεις, νέα νομοθεσία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Όταν κοιτάζω λοιπόν τα διάφορα θέματα τα οποία έθιξε, βλέπω ότι καταρχήν αναφέρεται στην κατάσταση του κοινοτικού δικαίου, της κοινοτικής νομοθεσίας και ε, βλέπουμε ότι σε ορισμένα θέματα είμαστε πολύ προηγμένοι σε σύγκριση με άλλες περιοχές και αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ζητήσει κανείς περισσότερη νομοθεσία. Μετά τη Λισαβόνα είμαστε ε, σε μία περίπτωση τρίτη φατίγκ είμαστε κουρασμένοι από τις συνθήκες Δηλαδή ε, δεν, ε, δεν, θέλει, ε, δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να υπάρξει μία αναθεώρηση των θεσμικών οργάνων. Από την άλλη πλευρά βρισκόμαστε στη θέση ότι έχουμε πάρα πολλές νομοθεσίες που δεν έχουν εφαρμοστεί και που δίνουν μεγάλες δυνατότητες για να επιλύσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε διότι αδιαφυσβήτητα μπορούμε στην Ευρώπη να πετύχουμε μακροπρόθεσμα μόνο ε, αν ε, ε, λύσουμε το θέμα της ενέργειας μακροπρόθεσμα και ό,τι και να σκεφτόμαστε για τις κλιματολογικές αλλαγές η αποτελεσματογικότητα της παραγωγής ενεργείας είναι πάντοτε πολιτικά ορθρό. Το CCF, το Carbon Capture and Storage είναι βασικό θέμα. Πρόκειται όμως για τεχνολογία που δεν χρειαζόμαστε ίσως. Η τεχνολογία υπάρχει στην αγορά κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η συνήθις τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι λογικό όσον αφορά τα δίκτυα, διότι μιλάμε μιλάμε πολύ ε, για την ανανεώσιμη ενέργεια αλλά χρειάζεται να αναπτύξουμε τα δίκτυα που υπάρχουν και πιστεύω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε ό,τι υπάρχει και δεύτερον τι καινούριο μπορούμε να δημιουργήσουμε. Διαφορετικά δεν θα ε, είμαστε αξιόπιστοι από τους πολίτες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να περιορίσουμε σε δύο λεπτά τις, ε, τις, ε, τα σχόλια. Ο Ζιλ με μεγάλη μας χαρά σας ε, καλωσορίσουμε εδώ, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, ο Τζο Λάινεν, και μαζί με τον Ζακ Ντελόρ ήμασταν μαζί πέρσι το Μάιο όταν διοργανώσατε αυτή την διάσκεψη για να δούμε κατά πόσο υπάρχει αυτή η κοινή θέληση αντιμετώπισης στο θέμα της ενέργειας. Και είδαμε και το σύνολο αυτού του σχεδίου μας ε, μιλήσατε για την εμβέλεια του προγράμματος και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική που εγώ υποστηρίζω ένθερμα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα εφαρμόσουμε τα οικονομικά αυτά σχέδια για την έρευνα και την ανάπτυξη, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε τον αντίστοιχο προϋπολογισμό ο οποίος να αφορά αποκλειστικά την ενέργεια. Στη συνέχεια, πώς θα πείσουμε για αυτή την συνδεσιμότητα, δηλαδή να έχουμε ευρωπαϊκά δίκτυα παρά μια πληθώρα εθνικών δικτύων που συνυπάρχουν. Και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πολύ στις ομαδοποιημένες αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτός είναι ένας από τους πολλαπλούς στόχους αυτής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας. Και σε σχέση με τον προλαλήσαντα θεωρώ ότι το άρθρο 294 της Νέας Συνθήκης είναι ανεπαρκές αν θέλουμε να φέρουμε εις πέρας αυτή την ε, πολιτική ενεργείας. Για να δούμε πώς ε, και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προβάλλουμε μια νέα πρωτοβουλία επί του θέματος. Άννα Ρόσπαχ. Er Σας ευχαριστώ πολύ γιατί προσήλθατε και σας ευχαριστώ γιατί επισκεφθήκατε και τη Σανγκάη. Θα ήθελα να σας πω τι πιστεύετε για το ε, Gazprom, για την Gazprom και το νέο αγωγό, ο οποίος δεν θα περάσει από την Πολωνία αλλά κάτω από τη Βαλτική. Επίσης, ως προς την Κίνα και τις ενεργειακές απαιτήσεις της ε, Κίνας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούν ε, μόνο άνθρακα ή περισσότερο άνθρακα και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι ως προς την ποιότητα του αέρα και της ατμόσφαιρας. Άρα ερευνούν και άλλες δυνατότητες, δηλαδή να αγοράσουν πετρέλαιο από το Ιράν το οποίο θα σημαίνει ότι θα αλλάξει και η πολιτική τους θέση ως προς το Ιρανικό πολιτικό σύστημα. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Θα πρέπει να κλείσω ε, τον κατάλογο μιλητών πλέον, λέει ο πρόεδρος. Πρόεδρε, Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μόλις ε, είπατε. Ένα μήνα πριν ήμουνα στην αντιπροσωπεία της Ινδίας, γιατί την προαναφέρατε. Βρεθήκαμε στο Νέο Δελχή, στο Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και συναντηθήκαμε για πάνω από μία ώρα με βουλευτές ε, Ινδούς που ενδιαφέρονταν για τις κλιματικές αλλαγές και ήταν πολύ καλύτερα πληροφορημένοι από μας διότι είχαν ε, μία εξειδίκευση, μία ειδίκευση επί του θέματος. Είχαμε μία ενθουσιώδη συζήτηση και στο τέλος ο επικεφαλής μας είπε ότι θα πρέπει να προβούμε στη σύσταση μιας κοινής επιτροπής για ανταλλαγές απόψεων. Και θεωρήσαμε ότι η ιδέα είναι εξαιρετική. Το πώς θα το κάνουμε είναι κάτι το διαφορετικό. Αλλά πώς σας φαίνεται η ιδέα καταρχήν. Και δεν ξέρω κατά πόσο στο Πεκίνο υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε μία κοινή μία, ένα φόρουμ τέλος πάντων για να το συζητήσουμε γιατί είναι το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουμε ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε, γιατί και εγώ σας έστειλα μία επιστολή εξ ονόματος της Επιτροπής ε, για την προστασία του κλίματος ε, και αυτό είναι ε, ένα θέμα, ένα ύψιστο αγαθό και αφορά όλες αυτές τις χώρες που προαναφέρθηκα. Η Λίντα Μαγκάβιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που έρχεστε παρόλο το βεβαρημένο πρόγραμμά σας ε, για να προωθήσετε ε, την εξοικονόμηση ενεργείας και την πρόθεση και βελτίωση του κλίματος. Αλλά όλοι έχουμε πάρα πολλή νομοθεσία. Δεν χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία. Αναρωτιέμαι όμως εάν προοδεύουν ε, τα κράτη ε, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Μετά, όσον αφορά την φθηνή ενέργεια, αυτό που χρειαζόμαστε είναι βιώσιμη ενέργεια, διότι ε, στην πρώτη προσπάθεια μειώσαμε τα ενεργειακά μέσα και βλέπετε οι Αμερικάνοι τώρα έχουν ε, να πληρώσουν το τίμημα της ελήψεως νομοθεσίας σχετικά με το πετρέλαιο και ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε σε συγκεκριμένα θέματα. Συμφωνώ με το Carbon Capture and Storage διότι η Επιτροπή έχει διαθέσει χρήματα για πιλωτικά προγράμματα αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να χρησιμοποιήσει κανείς τα χρήματα αυτά και ελπίζω ότι σαν πρόεδρος του Κοινοβουλίου ε, θα ασχοληθείτε με ε, το ίχνος άνθρακα ε, και μου είπαν όταν παραπονέθηκα ότι κάνει πολύ κρύο εδώ ότι υπάρχει κεντρικό air conditioning και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ενώ θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τα παράθυρά μας. Βλέπετε λοιπόν ότι τελικά θα κριθούμε από τα μέσα ενημέρωση από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο Κοινοβούλιο και από αυτού θα πρέπει επίσης κάτι να κάνουμε. Καλέσαμε τον κύριο Βέλε, ε, τον Γενικό Γραμματέα, να έρθει να μας πει ε, πώς διαχειρίζεται τα συστήματα. Ο Κρήτον Αρσένης. Ευχαριστώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που είσαστε εδώ, διότι πιστεύω ότι ο ρόλος σας για τα κλιματολογικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι πολύ σημαντικός. Θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπε η Λίντα Μακάβερν. Έχουμε ένα στόχο ε, μειώσεως 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε όμως πολύ περισσότερα. Ξέρω ότι η συμφωνία της ε, Κοπενχάγης δεν ε, επαρκεί για να αποφύγουμε τις κλιματολογικές αλλαγές και όπως ελέγχθη πρέπει να προχωρήσουμε σε μία μείωση 30% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εδώ στο Κοινοβούλιο με την ήμας έχουμε ήδη έναν στόχο του 30% ίσως όμως πρέπει να αυξήσουμε το στόχο αυτό. Ε, ε, σε αυτό το κτίριο παραδείγματος χάρη μπορούμε σε σχέση με την Ευρώπη να κάνουμε ε, πολύ περισσότερα και να δείξουμε ότι κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Μήπως μπορούμε λοιπόν να καθορίσουμε σαν στόχο ε, ε, ένα ε, carbon footprint ίχνος άνθρακα το οποίο να είναι της τάξης του 50% διότι διαπίστωσα ότι ορισμένες αίθουσες μένουν μένα τα φώτα όλη τη νύχτα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιες σπατάλες και πιστεύω ότι όταν οι πολίτες μαθαίνουν αυτά τα γεγονότα ε, ανησυχούν πάρα πολύ και ε, θα πρέπει να ε, βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Μάριο Πιρέλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτίμησα ιδιαίτερα και χτες και σήμερα την ε, παρουσία του Προέδρου Μπούζεκ. Ε, ιδιαίτερα επειδή προσέδωσε μεγάλη ε, προσοχή σε ζωτικά ζητήματα της καθημερινής μας ζωής. Νομίζω ότι πρόκειται για μία πρόταση η οποία πραγματικά είναι εξαιρετική. Ο κύριος Μπούζεκ ήταν ε, για πέντε χρόνια μέλος αυτής της Επιτροπής και εργάστηκε πολύ σκληρά. Συμφωνώ όταν μας λέει ότι μπορούμε να βγούμε από την οικονομική κρίση αναπτύσσοντας ε, εναλλακτικές ε, βιώσιμες και βιώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια. Χρειαζόμαστε έναν φορέα ο οποίος να ασχοληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ασχοληθεί με τη συρρήκνωση του κόστους. Να αποφύγουμε τις ε, σπατάλες και να προβούμε σε σωστό ενεργειακό εφοδιασμό. Μέσα στα πλαίσια μιας γενικής ε, αποταμιευτικής τάσης. Στη Βόρειο Ιταλία μία σχολή ασχολήθηκε ειδικά με αυτό το θέμα και προέβαλε ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να προταθεί και αλλού στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση της Ενέργειας και επ' αυτού θα ήθελα να σας υποβάλω τις εξής ερωτήσεις. Τι δυσκολίες υπάρχουν για να υπάρξει αλληλοκατανόηση μεταξύ των 27 κρατών μελών και ε, ποιος θα ήταν ε, ο χρόνος υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να σας διακόψω. Ο Πίτερ Λίζε. Μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ, Πίτερ Λίζε. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητέ Γέρζη που επιστρέφει στη βαλιά σου επιτροπή. Έχω ε, δύο ερωτήσεις και παρατηρήσεις για την Κίνα. Πρώτον, θα πρέπει να προσέξουμε σε άλλες αναδυόμενες χώρες να μην τις βάλουμε όλες στο ίδιο τσουβάλι με την Κίνα. Για μένα οι χώρες ε, που είναι πιο θετικές στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και υποστηρίζουν τη διαδικασία χρειάζονται και τη δική μας υποστήριξη για να ασκήσουμε από κοινού πίεση στην Κίνα και στις Ηνωμένες και στην Κοπεχάγη πάλι διχάστηκε ο κόσμος ε, η βιομηχανικά κράτη και οι υπόλοιποι μαζί με την Κίνα. Και η Κίνα ε, προσετερίστηκε και το Μεξικό και τη Βραζιλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την προστασία του κλίματο, αλλά και για την μελλοντική παγκόσμια τάξη. Γιατί οι συγκρούσει. Ε, συμφερόντων που έχουμε δεν είναι όλες οι κοινές ε, των χωρών αυτών απέναντί μας. Πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Eurolat με τους συναδέλφους από τη Λατινική Αμερική και ακούσαμε ε, άλλα πράγματα από αυτά που λέει η Κίνα. Θέλουν πάρα πολύ να πετύχει η διαπραγμάτευση στη Κανκούν ή το αργότερο στη Νότια Αφρική και θα πρέπει και εμεί να το υποστηρίξουμε. Με Βραζιλία, Μεξικό, Νότια Αφρική, μαζί από κοινού να ασκήσουμε πίεση στην Κίνα και μου έκαναν εκεί μια πρόταση, τη διαβίβασα και στον πρόεδρό μας, τον Γιώ Λάινεν, γιατί να μην στείλουμε αντιπροσωπεία από χώρε όπω είναι το Μεξικό, η εκπρόσωπο του Μεξικού το υπέβαλε αυτό, στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Κίνα. Δηλαδή, να λέμε τα κοινοβούλια των χωρών που έχουν δέσμευση και προσήλωση για διεθνεί συμβάσει, ε, από κοινού λοιπόν να εργαστούμε και να επισκεφθούμε και την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Το άλλο δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, αλλά με την έκθεση Ανδρέ Περίγιο που εγκρίναμε την περασμένη φορά στην Ολομέλεια. Μιλήσαμε για αυτό το αποτρόπαιο ε, έγκλημα που γίνεται ε, θανάτωσης με σκοπό την αποκόμιση των ε, οργάνων των ανθρώπων. Θα το θέσεις υπόψη των Κινέζων αυτό, ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι διανύουμε μία πολύ ε, σημαντική χρονική περίοδο και εγώ ήμουνα στην ε, Κίνα και ήρθα σε επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος μας είπε ότι κλείνουν οι μονάδες παραγωγής άνθρακα, ιδιαίτερα αυτές οι μονάδες οι οποίες είναι απαρχαιωμένες, διότι θα ε, μπορούσαν να διπλασιαστούν σε σχέση με τις παλές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό τουλάχιστον κλείνουν οι πιο παροχημένες. παροχημένες. Στην Ευρώπη δεν έχουν γίνει τέτοιε συζητήσει. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς μπορούμε να ξαναμπούμε σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή να προβάλλουμε νέε προτάσεις σε σχέση με τον έλεγχο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Εμείς δεν έχουμε ε, συμμετάσχει ενεργά και ούτε το κάναμε στη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικά σοβαροί, νομίζω ότι μπορούμε να προβάλλουμε ένα άμεσο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα κρούσης για ε, να μετακινηθούμε από τη, την, την ενέργεια ορυκτών καυσίμων στις ανανεώσιμες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το, το ευκταίο και το εφικτό έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και την συγκυρία. Δηλαδή, αν θέλετε να αναποδογυρίσουμε, να αντιστρέψουμε τη συγκυρία. Θα πρέπει αυτό ακριβώς να κάνουμε και πολύ σοβαρά και αυτό σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η πραγματική ε, πρόκληση και το κρίσιμο σημείο μεταστροφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που βρίσκεστε μαζί μας. Αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια στιγμή κρίσης και οικονομικής και ενεργειακής και περιβαλλοντικής σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που χρειαζόμαστε φυσικά είναι γενναίε πολιτικές, που εμείς λέμε πράσινες πολιτικές. Να σημειώσουμε ότι αυτή η συζήτηση για την Κίνα είναι λίγο υποκριτική γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκά συμφέροντα και σε σχέση με, τα, με τον διεθνή καταμερισμό. Εμείς χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Συζητάμε για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με μείωση 40% ως το 2020 των αερίων παράγων του φαινόμενου του θερμοκηπίου. 80% μέχρι το 2050. Χρειαζόμαστε απεξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια και όχι από την πίσω πόρτα υποστήριξή της. Και μάλιστα στη Μεσόγειο αυτό μας ενδιαφέρει με τα καινούργια πυρηνικά προγράμματα της Τουρκίας. Χρειαζόμαστε έμφαση στην, στην εξοικονόμηση ενέργειας που είναι μια τεράστια πηγή και φυσικά η πολυευρωπαϊκή πολιτική σε μεγάλο βαθμό είναι κενό, κενά λόγια. Χρειαζόμαστε επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, στις μεταφορές και στις κατασκευές. Ο πράσινος στόχος για τις ανανεώσιμες μέχρι το 2050 είναι 100%. Χρειαζόμαστε ανανεώσιμες μορφέ μορφές στις μεταφορές με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αξιοποίηση των υπολοιμάτων της αγροτικής και της δασικής βιομάζας. Μιλάμε για νέες τεχνολογίες. Ναι, Βεβαίως, μιλάμε και για έξυπνα δίκτυα στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά βεβαίως. Αυτό όμω που κυρίω χρειαζόμαστε είναι η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξη, που οι κυρίαρχες δυνάμεις έχουν επιβάλει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και του μοντέλου κατανάλωσης. Ο απλό πολίτη δεν είναι έξω από το στόχο. Γι' αυτό και ζητούμε να αλλάξουν οι πολιτικέ, να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπίε αλλά πάνω απ' όλα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναποκτήσουμε έναν ρόλο πρωτοποριακό που είχαμε στο παρελθόν και φάνηκε να χάνουμε το βηματισμό μας. Ευχαριστώ. Ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο που μίλησε για την κατασπατάληση ενέργειας με τον κλιματισμό ε, εδώ και στο Στρασβούργο. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο ε, Μπούζεκ για την αφήγηση αυτή, για την παρουσίαση δηλαδή, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ειδικό βάρος επί του θέματος. Ως προς την ε, Κίνα, είναι σαφές ότι η Κίνα τα επόμενα χρόνια θα μειώσει την κατανάλωση και παραγωγή του άνθρακα, άρα θα επιβαρύνει κατά πολύ την ατμόσφαιρα. Επίσης, δεν πρέπει να κάνουμε δώρα στην ε, Κίνα τη στιγμή που εμείς καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες και στην ουσία επιβάλαμε φόρους σε χώρες που κάνουν εισαγωγέ που δεν τηρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό δεν το κάναμε για την Κίνα. Τι γνώμη έχετε, θεωρείτε ότι ε, δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε φόρους και στους μεγάλους παραγωγούς ε, άνθρακα. Σε σχέση με αυτά που προείπατε, δεν ξέρω κατά πόσο ε, θα πρέπει οι κλιματικές αλλαγές να επιβαρύνουν αποκλειστικά την Ευρώπη. Ενώ εμείς καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες και θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες οικονομικές προσπάθειες από τρίτες χώρες που είναι μεγάλοι μολυντές. Γιατί δυστυχώς το έγγραφο το οποίο βγήκε από αυτή την αίθουσα, από την Ολομέλεια και έφτασε στη Κοπενχάγη μίλησε υπέρ τρίτων χωρών χωρίς να ζητήσουμε ένα αντιστάθμιο από τις χώρες αυτές που είναι οι μεγάλοι μολυντές της φιλίου. Ευχαριστώ κυρία Κάλαμπαχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για την Κίνα, τα πυρηνικά εργοστάσια και τις ε, πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Και θα ήθελα να σας μιλήσω για το Μοχόφσκ που είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο στα 160 χιλιόμετρα από τη Βιέννη και όχι τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες αλλά τεχνολογία της δεκαετία του 70. Έχει συμμετάσχει ε, και από την Αυστρία σε διαμαρτυρίες πολιτών εκατομμύρια κατά τις ε, διαδικασίες αυτής που είναι στο στάδιο 3 και 4 και καταλαβαίνετε ότι ε, παραβιάζονται από τις σλοβακικές αρχές ε, οι τα δικαιώματα των ε, πολιτών μας και της χώρας μας και της Κάτω Αυστρίας και της Άνω Αυστρίας στα διάφορα κρατήδια έχουμε απευθυνθεί στον αρμόδιο επίτροπο Έτιγκερ και όπου δει αλλά θα παρακαλούσαμε ε, και εσείς ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας υποστηρίξετε γιατί και εμείς έχουμε ε, ως Κοινοβούλιο ψηφίσει αυτή την οδηγία και να προωθήσουμε στην Ευρώπη μαζί σας την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas prezidentė, labai malonu, kad jūs... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας ε, σχετικά με τα ενεργειακά δίκτυα τα οποία αναπτύσσονται εις την Βόρειο Θάλασσα. Εκεί βέβαια υπάρχουν ορισμένοι πολιτικοί περιορισμοί και περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στο carbon capture and storage ή στην αιωλική ενέργεια τα οποία πρέπει να προωθήσουμε αλλά και άλλες ε, πηγές ενεργείας και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας σχετικά με το πώς μπορούμε να ε, κάνουμε μία ανεξάρτητη ε, μελέτη των επιπτώσεων κατά τρόπον ώστε τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται εις ε, τις παράκτιες χώρες της Βορείου Θαλάσσης και στις ε, ε, χώρες που παραμεθορίως χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να απαντήσετε σε όλα αυτά σε πέντε λεπτά αλλά τουλάχιστον πέστε μας τι είναι βασικό. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Να σας απαντήσω γενικά ή πιο εξειδικευμένα, πιο συγκεκριμένα. Θα προσπαθήσω να ε, σας απαντήσω αφιερώνοντας 20 δευτερόλεπτα στον καθένα. Το πολύ 30. Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ο χρόνος. Ε, προς τον πρώτο συνάδελφο. New rules. We have in Lisbon Treaty. Προς τον συνάδελφο Ζέμπερ. Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας για την ελληνική στον ενεργειακό τομέα. Η ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά δεν έχει εγγραφεί έτσι στη συνθήκη. Πρόκειται για ένα διαθεσμικό ζήτημα. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια Τίποτα δεν έχει ε, εγγραφεί επακριβώς έτσι στη συνθήκη. Εμείς θα πρέπει να βρούμε την ε, ουσιαστική λύση. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Θα πρέπει να εκπληρώσουμε ε, το, το γράμμα της συνθήκης, αλλά ευρύτερα, πολύ ευρύτερα από ό,τι καταγράφεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Σε τρία, τέσσερα, πέντε σημεία. Ενέργεια, κλιματικό ζήτημα. Και αυτό σχετίζεται με το δικό σας ε, ερώτημα, το οποίο είναι ε, μεγάλη σημασία. Κύριε Πανιό, έχετε δίκιο. Βεβαίως, το χρηματικό είναι το βασικό. Εμείς θα αποφασίσουμε για τον επόμενο προϋπολογισμό πόσα χρήματα θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Όχι να πούμε ότι μετά τον προϋπολογισμό, την κατάρτισή του, α, χρειαζόμαστε και κάτι για την ενέργεια, για τα ενεργειακά δίκτυα, για τις κλιματικές αλλαγές και, και, και. Θα πρέπει να το ορίσουμε τώρα. Ναι ή όχι. Ή ας πούμε όχι, αν δεν θέλουμε. Όλα εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Αυτόν πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου. Ως προς την ενιαία αγορά, τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, ήταν μια ιστορία μεγάλης, μεγάλων επιτυχιών. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έπρεπε να προετοιμάσουν το νομοθετικό έργο, αλλά τα κράτη-μέλη επιθυμούσαν την ενιαία αγορά. Αυτό πρέπει να συζητήθει με τα κράτη-μέλη. Μετά τη συζήτησή μας ε, εδώ θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα για την ζωτικής ε, σημασία. Με την υποστήριξη βεβαίω των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Χωρίς τη δική σας υποστήριξη ε, θα είναι νεκρό γράμμα αυτή η ιδέα. Και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα, τα ενεργειακά κοινής έρευνας. Θέλουμε χαμηλού κόστους ενέργεια, μα δεν μπορεί να γίνει χωρίς ε, τις ανανεώσιμες, χωρίς την ε, βελτίωση των τεχνολογιών, γιατί είναι ιδιαίτερα δαπανηρές οι τεχνολογίες. Θέλουμε να κάνουμε επιμερισμό των δαπανών ή όχι. Ή κάθε κράτος μέλος θα κινηθεί ξεχωριστά. Ξέρουμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έχουμε το 7ο και θα έχουμε σύντομα το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό είναι προστιθέμενη αξία. Θέλουμε να το επιτύχουμε και στον ενεργειακό τομέα, ναι ή όχι. Άρα ε, βρισκόμαστε στην απαρχή των συζητήσεων. Δύο μέρες πριν ε, συζήτησα το θέμα στην Επιτροπή Ήτρε. Τώρα το συζητώ δεύτερη φορά με εσά. Είναι μια πολιτική ιδέα. Εν το γίγνεστε. Μιλώντας για την Κίνα λοιπόν, υπήρξε και μία άλλη ερώτηση, πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, του CCS και συνεργασία με Κίνα και Ιράν. Δεν συζήτησα ένα τόσο εξειδικευμένο ζήτημα ως προς τη συνεργασία της Κίνας με άλλες χώρες ανά τον κόσμο ιδιαίτερα ως προς την ε, παροχή, την προμήθεια πετρελαίου. Βεβαίως συζητήσαμε για το Ιράν από πλευράς ασφάλειας και η Κίνα θα υποστηρίξει τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως ξέρετε, έστω και αργά. Δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά το συζητήσαμε επακριβώς με τις κινέζικες αρχές, αλλά όχι σε συσχετισμό με θέματα εφοδιασμού ενέργειας. Αυτό ήταν κάτι το διαφορετικό. Αυτά ως προς τη σχέση Κίνας-Ιράν. Ως προς την Ινδία. Εξαιρετική η ιδέα σας. Στην ε, περίπτωση είπα η Ινδίας και η ΜΟΝ. Έχουμε μια κοινή επιτροπή. Βεβαίω θα την υποστηρίξω όποτε θέλετε. Αλλά με την Κίνα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα γιατί θα ήταν πολύ καλό να υπάρχει μια τέτοια κοινή επιτροπή, αλλά δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις, είναι κάπως διαφορετικό το ζήτημα. Δεν θέλω να πω όχι, γιατί θα ήταν σημαντική συνεργασία, αλλά στην Ινδία υπάρχει δημοκρατία. Πρόκειται για μια τεράστια χώρα, η οποία ε, είναι μια μεγάλη δημοκρατία, μεγαλύτερη δημοκρατία ανά τον κόσμο. Άρα την υποστηρίζω αυτή την ιδέα και σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακέβαν ε, υπέβαλε μια ερώτηση. Συμφωνώ με αυτά που προείπατε για τις διαπραγματεύσεις, για την εκστρατεία αυτή, τη γενικότερη, πώς μπορούμε να επικεντρώσουμε τους στόχους μας, να μιλήσουμε για τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να ε, πούμε ειλικρινά ότι Είχαμε υψηλές προσδοκίες από την Κοπενχάγη. Εδώ μιλάμε για ένα κατόφλι σε σχέση με το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Όμως, ας κρατήσουμε το ρυθμό των συζητήσεων για να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε στο Κανκούν. Πολύ συνεργαζόμαστε επ' αυτού. Και μπορώ να σας πω ότι και πάλι θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολα τα επόμενα βήματα, αλλά θα πρέπει να κατέχουμε ηγετική θέση. Και όπως είπε και ο Πίτερ Λίζε, λίγα λεπτά πριν, αυτό θα πρέπει να γίνει μαζί με άλλους. Αναπτυσσόμενες ε, χώρες, αναδιόμενες, οικονομικά χώρες, δηλαδή μην κατακαιρματίζουμε τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος μας πριν τις διαπραγματεύσεις, να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς, με τους Κινέζους. Δεν θέλουν να υπογράφουν δεσμευτικές ε, συνθήκες, το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Χωρίς δεσμευτικές συμφωνίες δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα ας επιλύσουμε ορισμένα ζωτικά ζητήματα, δηλαδή τα, τα ταμεία προσαρμογής, δηλαδή να υποστηρίξουμε την προσαρμογή, τη σταδιακή προσαρμογή, ιδιαίτερα για τις αναδιόμενες ε, χώρες, διότι φαίνεται ότι αυτά τα ζητήματα είναι ξεχωριστά, αλλά είναι αλληλένδετα. Και ως προς τη ροή της τεχνολογίας. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή, ποιοι είναι οι κανόνες τεχνολογία, ε, προσαρμογή Όλα αυτά αποτελούν ψηφίδες του συνόλου, διότι χωρίς αυτές τις μικροσυμφωνίες δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην τελική δεσμευτική συμφωνία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και η κυρία Χάτιγκαρτ, η οποία μας εκπροσωπεί, μας εκπροσωπεί πάρα πολύ καλά. και δεν είναι και τόσο αισιόδοξη πολλές φορές. Άρα ούτε και εγώ. Άντε, ας πούμε 90%. Ως προς το αποτύπωμά μας και το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Γνωρίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και το CCS και για το στόχο του 20% που αναφέρθηκε. Ίσως μετά την παρέμβασή σας ε, θα μπορούσα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα πέμπτο σημείο της ενεργειακής πολιτικής. Να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Αυτό. Εντάξει, το άνοιγμα των παραθύρων, ας πούμε. Και αυτό, κάτι είναι και αυτό. Τις γενικές μας συνήθειες. Πώς να κινούμαστε στις ΠΟΠ στις πόλεις με ποδήλατο. Άρα ίσως το πέμπτο σημείο θα έπρεπε να είναι στην πρότασή μου αυτό. Γιατί σας μίλησα για την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας, την δικτύωση, το Ταμείο Ενέργειας για τις ε, τεχνολογίες και τις επιχειρήσεις προμηθειών. Πέμπτο λοιπόν, αλλαγή των συνηθιών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Το επόμενο ερώτημα αφορούσε τις ε, κλιματικές αλλαγές και τα κράτη-μέλη. Βεβαίως όλα εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή μας ε, Ένωση. Πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι στις ε, αποφάσεις μας μέσω των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, των Συμβουλίων Υπουργών και μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι ένας νέος θεσμός. Άρα αυτό θα πρέπει να το προωθήσει και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Βαν Ρομπόη. Όπως είπε και η κυρία Μακέβαν, χωρίς την υποστήριξη των κρατών μελών δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι ο απότερος στόχος. 20 ή 30% στο μέλλον. Ο Πίτερ Λίζε υπέβαλε ένα ερώτημα σε σχέση με το τι λένε οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι λένε είμαστε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Δεν είμαστε αναπτυγμένη χώρα. Άρα χρειαζόμαστε υποστήριξη. Άρα δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε τις ε, εκπομπές. Θα περιμένουμε έτσι ώστε οι εκπομπές, οι κατακεφαλή εκπομπές να είναι ίδιες με τις δικές σας χώρες. Αυτό σημαίνει σε 10-20 χρόνια. Είμαστε μία αναδυόμενη χώρα. Δείτε τα στατιστικά στοιχεία. Άρα η συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσβατη για το ζήτημα αυτό. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους Κινές, όπως είπε ο Πίτερ Λίζε. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό στην Κίνα. Το αναφέρω κάθε φορά και το δέχομαι και το συζητώ με τους υπουργούς Μιλώ για θέματα ενέργειας, κλιματικών αλλαγών και άλλα συναφή. Θα βρεθώ στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα τους ε, μιλήσω για τις συνομιλίες μας, διότι βεβαίως έχει μεγάλη σημασία για την, έχει μεγάλη σημασία για την υποεπιτροπή αυτή. Ο Βιτόριο υπέβαλε ένα ε, ερώτημα το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ένα πιο επιθετικό πρόγραμμα με την Κίνα, έναντι της Κίνας. Με, με Βιτόριο, φαίνεται ότι σε ενόχλησα μπορούμε να συζητάμε για άλλους στόχους και για την ε, ανάπτυξη των ανανεωσίμων. Αυτό αφορά την ε, ασφάλεια προμηθειών. Δεν αφορά μόνο το κλιματικό. Και είναι πολύ δύσκολο να το συζητήσουμε με τους Κινέζους. Μόνο αν τους ε, παρέχουμε δωρεάν τεχνολογία μπορεί να γίνει αυτό. Αν τους δώσουμε τεχνολογία του CCS, δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι αποδοτικό κάτι τέτοιο, πρέπει να το ελέγξουμε πρώτα στην Ευρώπη. Και ένας συνάδελφος είπε ότι δεν μπορούμε να τους δώσουμε, να τους παρέχουμε τεχνολογία δωρεάν και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Εάν θέλουμε να τους δώσουμε, να προβάλλουμε μία δωρεάν παροχή του CCS ή των ανανεωσίμων, της αποδοτικότητας των τεχνολογιών και ούτω καθεξής ή όχι. Έχει μεγάλη σημασία η αποδοτικότητα κατά την παραγωγή ενέργειας. Αυτό αφορά και τις μονάδες παραγωγής άνθρακα γιατί μπορεί η αποδοτικότητα να είναι 35 ή 50, 60%. Εάν συνδυαστεί με ε, ένα πρόγραμμα της ε, παραγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου διότι είναι μεγάλη η αποδοτικότητα, θα μπορέσουμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε ε, την τεχνολογία μας. Γι' αυτό και Βιτόριο, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα οποία είπε, ήταν πολύ σημαντικά έγινε και μία ερώτηση από ε, τον ε, κύριο Τρεμόπουλο. Με συγχωρείτε δεν γνωρίζω το όνομά σας αλλά θα το μάθω σχετικά με ε, τα ε, δίκτυα είναι πολύ βασικό θέμα. Ε, πρέπει να λύσουμε ορισμένα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κονδύλια για την τεχνολογική πρόοδο. Χρειαζόμαστε δηλαδή πόρους και ε, επίσης ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, τις προτάσεις σας που δίνουν στην Ευρώπη μία προστιθέμενη αξία. Μοναδικό πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Πολύ σωστά. Για κύριε Ρώση, ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Μιλήσατε για την Κίνα. Αν θα είναι δώρο ή θα τους πουλήσουμε την τεχνολογία θα εξαρτηθεί από την αντιμετώπιση τους του προβλήματος. Γιατί λέγουν είμαστε μια υποανάπτυξη ε, χώρα, άρα δεν χρειάζεται να μειώσουμε πολύ τις εκπομπές μας. Διότι θα θέλαμε να αναπτύξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά βεβαίως υπάρχει και το πρόβλημα της ρυθμίσεως στον ΠΟΕ στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου για ε, την φορολόγηση του διεξιδίου του άνθρακος. Ε, αυτό είναι μία πρόταση των Γάλλων για τα σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η κυρία Κάλεμπαχ Αναφερθήκατε στα πυρηνικά θέματα. Η αντιμετώπιση είναι διαφορετική αναλόγως των κρατών μελών, άρα είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Ξέρω ότι υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των χωρών που ήταν πολύ σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Και τέλος, και επίσης σημαντικό, η Βαλτική ε, εδώ αναφερόμαστε στην ε, ευρωπαϊκή ενεργειακή μας κοινότητα. Σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, ε, νότιο-ανατολικά, νότιο-δυτικά, και εχωμένος ε, στην ε, ε, κεντρική ανατολική πλευρά της Ευρώπης υπάρχουν απομονωμένες νησίδες που χρειάζονται μία δημιουργία δικτύου, μία στήριξη για ανανεώσιμες νέες τεχνολογίες σε όλες τις χώρες και όχι μόνο σε αυτές που προανέφερα. Οπότε, σε ορισμένες χώρες νομίζω ότι τώρα αναμφισβήτητα τα προγράμματα αυτά είναι πολύ θετικά και όλα στο τέλος εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη και από τη στήριξή τους. Κάθε συζήτηση την οποία διεξάγω στις χώρες στις οποίες έχω επισκεφτεί επισήμως και είναι 14 χώρες ε, μέλη της ε, ενεργειακής κοινότητας της Ευρώπης όπου μιλάμε για συγκεκριμένη δικτύωση χρηματοδότηση της έρευνας ε, πουθενά δεν υπήρξε ανητική αντίδραση όλοι είπαν θα το δούμε είναι καλή ιδέα αλλά πρέπει πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον. Χρειάζομαι στήριξη. Όλοι μας χρειαζόμαστε στήριξη. Και από τα εθνικά κοινοβούλια και ακόμη και αν συμφωνούμε με αυτή την ε, γενική ιδέα πρέπει να προωθήσουμε το πρόγραμμα αυτά. Εμείς πρέπει να την προωθήσουμε διότι δεν είναι κανείς έτοιμος και εμείς δεύτερη συζήτηση κάνουμε μόνο επί του θέματος αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για την ε, υπομονή τους γιατί ξεπέρασαν την ώρα τους 10 λεπτά. Δεν ήμουν τόσο σύντομος ε, όσο ήλπιζα, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με τα χαράς ε, ε, βλέπω ότι είσαστε πολύ προσιλωμένος στα θέματά μας και θα δεθεί το μήνυμα προς όλα τα μέλη της Επιτροπής μας ότι είσαστε προστηλωμένος στους στόχους μας και λίγεται η συνεδρίαση. Η επόμενή μας συνεδρίαση είναι στις 21 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ.